Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Because we have quite a... Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε γιατί είναι βεβαρημένη η μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να σα σας καλωσορίσω όλους. Ξεκινάω αμέσω με το σημείο 1, την έγκριση της μερίσιας διάταξής μας. Αν δεν υπάρχουν ε, προτάσεις για μεταβολές, μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνεται Δεύτερο θέμα, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 3 και 4 Νοεμβρίου. Θα σας έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά και θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν έχετε αντίρρηση μέχρι το τέλος των συνεδριάσεων μας. Τρία, ανακοινώσεις της Προέδρου θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά επειδή έχουμε συνεδρίαση με τους συντονιστές αργότερα το απόγευμα, θα κάνω τις ανακοινώσεις μου αύριο, αν δεν έχετε αντίρρηση, και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 4, ανταλλαγή απόψεων με τον Κλάους Κλιπ. Παρακαλώ, ο Λόμπερ ζητά το λόγο. Μία ενημέρωση, πολύ σύντομη για την εξέλιξη μιας έκθεσης που ψηφίσαμε σε αυτή την Επιτροπή. Θέλω να πω πώς είναι η διαδικασία τώρα. Η πρότασή μας επανεξετάζεται στο Συμβούλιο και θέλουν να μεταβάλουν ορισμένα πράγματα. Είχαμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες που άλλαζε το την κατάληξη του κανονισμού και χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο από όσο ανέμενα για να έλθουν με μία πρόταση. Χθε μου δόθηκε η πρόταση. Σήμερα το πρωί είχαμε τρίλογο και καταλήξαμε σε συμφωνία με μικρομεταβολές. Όμως, και αυτό είναι το κέριο σημείο που θα ήθελα να σας αναφέρω, τώρα είμαστε κάτω από τη συνθήκη της Λισαβόνας και σημαίνει ότι μπαίνουμε σε αυτή τη νέα φάση που το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να έχει αυτή την περίοδο των 8 εβδομάδων για να αποφανθεί αν είναι θέμα επικουρικότητας ή όχι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τελειώσαμε την εργασία μας, αλλά πρέπει να περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Μάρτιο, προτού ληφθεί η απόφαση στην Ολομέλεια. Σας το εξηγώ λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, χαίρομαι πάρα πολύ που καταλήξαμε γι' αυτό, αλλά βεβαίως Παρόλο που είμαι ευτυχής είμαι και απογοητευμένος λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας που δεν μπορούμε να επισπεύσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νόμπερ, αυτό είναι ενημέρωση, δεν αφορά την ημερήσια διάταξή μας, αλλά θα αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερα προβλήματα το δεύτερο κανονισμό. Ευχαριστώ για την ενημέρωση πάντως. Άλλα σχόλια δεν υπάρχουν. Περνάμε στο 4 ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης. Καλωσορίζω τον Κλάους Κλίμπ, της ε, Γενικό Γραμματέα της συνέλευσης αυτής, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης έχει κάπου ιστορία 25 ετών ήδη και ο πιο ανεξάρτητος οργανισμός περιφερειών σε μια ευρύτερη Ευρώπη, δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 70 περιοχές που έρχονται από 33 χώρες και πολλούς περιφερειακούς φορείς και καλέσαμε τον κύριο Κλάους Κλίμπ για να μας ενημερώσει σχετικά με τις εργασίες της συνέλευσης, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της νέας συνθήκης και, και της πολιτικής συνοχής της Ευρώπης. Λοιπόν, δίνω απευθείας το λόγο στον Κλάους Κλίμπ και στη συνέχεια θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων βεβαίως. Κλάους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που ο πρόεδρος μας δεν μπόρεσε να έρθει. Στην Γαλλία έχει ξεκινήσει μια εκλογική καμπάνια για τις εκλογές της περιφέρειας και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Όταν έφτασα στις Βρυξέλλες χθες και ε, είδα ένα μεγάλο πλακάτ 1η Δεκεμβρίου είναι η μέρα για το AIDS. Αλλά ξέρουμε ότι είναι και η μέρα που τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Το 2002 ξεκίνησε η συνέλευση για αυτό το θέμα και τότε αν θέλετε μπήκα και εγώ στη συνέλευση των περιφερειών και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι στενά συνδεδεμένη με τις εργασίες μας στη συνέλευση των περιφερειών. Νομίζω ότι την επηρεάσαμε αρκετά. Τώρα ξέρετε ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας πραγματικά υπάρχει μια νέα αναγνώριση της επικουρικότητας του ρόλου των περιφερειών κτλ. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που βλέπω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς δηλαδή, έχετε αποκτήσει πραγματικά όλες τις εξουσίες ενός νομοθετικού σώματος. Αυτό είναι μια απαρχή καλής συνεργασίας μεταξύ ευρωβουλευτών και εκλεγμένων ηθινόντων στις περιφέρειες. Όπως είπε η Ντανούντα, η συνέλευσή μας συστάθηκε το 85. Έχουμε μέλη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. 30% λοιπόν είναι εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνεται και η Σουηδία και τα υπόλοιπα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και 16 οργανώσεις που είναι μέλη, όπως η Ένωση ε, Παραμεθόριων Περιοχών, ε- η Ένωση των Πυρηναίων, που θα μετατραπεί σε κάτι άλλο τώρα και κτλ. Η συνέλευση τι κάνει βασικά. Έχουμε δύο κλάδους. Λόμπινγκ είναι το ένα προς τα θεσμικά όργανα των Βρυξενόλ. Αλλά ακόμη και προς υποστήριξη των τοπικών μας φορέων στις συναλλαγές τους με τις κυβερνήσεις. Το άλλο κομμάτι είναι η πρακτική συνεργασία. Μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε σε, κάτω από τρεις του τίτλους, ανταλλαγή εμπειριών. Έχουμε μεγάλο εύρος μεθοδολογιών που χρησιμοποιούμε. Τις αναπτύξαμε μόνοι μας, χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία εμπειρογνωμένων από περιφέρειες. Έχουμε ανταλλαγή συναδέλφων, ε, ε, κατάρτιση, ε, διαγωνισμούς που τους χρησιμοποιούμε όχι για να δώσουμε κάποιο βραβείο, αλλά για να ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει σε ανάλογη περίπτωση σε περιφέρειες. Τώρα, στην πρακτική συνεργασία ασχολούμεθα με την ανταλλαγή εμπειριών. Έχουμε και πρόγραμμα επισκέψεων επαγγελματικών μετά την επαγγελματική κατάρτιση φοιτητών. Έχουμε και κάποια προγράμματα τα οποία επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ηγούμεθα τέτοιων σχεδίων, είτε συμμετέχουμε το 90% του προϋπολογισμού μας προέρχεται από την εισφορά των μελών και καμιά φορά έχουμε και επιδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη μας είναι μέλη διότι διάλεξαν να γίνουν μέλη και πληρώνουν εισφορά. Έχουμε μεγάλη αύξηση των εισφορών τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται αυτή η αυξητική τάση. Αυτοί είναι οι δύο τομείς λοιπόν ενασχόλησής μας. Τεχνικά ε, μοιραζόμαστε σε τρεις επιτροπές και δύο μόνιμες επιτροπές την Επιτροπή Οικονομίας και Περιφερειακής Πολιτικής, η δεύτερη είναι Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας και η τρίτη είναι για την παιδεία, την νεολαία και τον πολιτισμό. Θεσμικά θέματα ε, καλύπτονται από μόνιμη επιτροπή και το ίδιο ισχύει και για τις ίσες ευκαιρίες. Η συνέλευση των περιφερειών δεν είναι γραφειοκρατικό όργανο. Νομικά είμαστε μια ένωση. Δεν είμαστε μονόδρομος. Δεν έρχονται τα μέλη σε εμά για να μας πούνε κάτι. Είναι πραγματικά ένα ζωντανό δίκτυο στο οποίο τα μέλη μας είναι δραστήρια, δεν πληρώνουν απλώ συμμετοχή. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να οργανώσουμε συναντήσεις, ε, στις διάφορες περιφέρειες και ε, προγράμματα κατάρτισης, αλλά και οι περιφέρειες ε, έχουν τη δικιά τους τη δράση, συντάσσουν εκθέσεις, οργανώνουν διασκέψεις, συναντήσεις, καταρτήσεις. Είναι κάτι αρκετά μοναδικό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να σας πω, μέσω της συνέλευσης αυτής. Δηλαδή βρισκόμαστε παντού σε όλη την Ευρώπη σε 270 περιφέρειες. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, ας ξεκινήσω να σας λέω τι είδου Ευρώπη θέλουμε. Μια Ευρώπη που να παράγουμε ένα κανονισμό μετά τον άλλο ή θέλουμε μια Ευρώπη που να κινείται πραγματικά από τους πολίτες, από τις περιφέρειες. Θέλουμε μια Ευρώπη που να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις περιφέρειες να προχωρήσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναπτυχθούν. Μπορώ να συγκρίνω καταστάσεις σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης σαν να πετούσαμε από ελικόπτερο. Αν το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι αν συγκρίνετε τις περιφέρειες έτσι, ε, κάποιες είναι συγκρίσιμες, κάποιες μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά και σε 20 χρόνια έχουν προχωρήσει ουσιαστικά και άλλες περιοχές, άλλες περιφέρειες δεν, δεν προχωρούν ποτέ. Και πολλά μπορούν να γίνουν με αλληλεγγύη μεταξύ περιφερειών αλλά και με τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων. Η εκλεγμένη πολιτική της Ευρώπης όπως σας έλεγα, έχουμε μέλη από 33 χώρες, 33 διαφορετικά συστήματα οργάνωσης των περιφερειών συνεπώς. Αυτό που ενώνει τους ανθρώπους είναι οι εκλεγμένοι που πρέπει να καταφέρουν να πετύχουν για να ξαναεκλεγούν. Και έχουν τέσσερα χρόνια μόνο ε, συνήθως εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην οτροπία. Δεν υπάρχει δηλαδή επιλογή, είτε έχουν τους πόρους και τις δυνατότητες, είτε όχι. Πρέπει να προχωρήσουν και το πραγματοποιούν. Κάτι άλλο που μας διασυνδέει στενά με τους ευρωβουλευτές που είναι και αυτοί εκλεγμένοι είναι το εξής. Κάναμε μία μελέτη για την οικονομία και την κρίση τη δημοσιονομική την Άνοιξη. Όταν λοιπόν κάνετε μια τέτοια μελέτη, θα δείτε ότι έχουμε 22 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που αντιπροσωπούν αντιπροσωπεύουν 98-99% όλων των εταιριών της Ευρώπης και ε, προσφέρουν τα δύο τρίτα της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τα ξέρετε πιθανότατα αυτά, αλλά αυτά θέλω να το τονίσω και πάλι. Με μια τέτοια κρίση σαν και αυτή που έχουμε είχαμε, Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτές τις πολλές επιχειρήσεις που μπορεί να χρεοκοπήσουν. Εάν έρθετε σε επαφή με 5 ή 10% μιλάτε 100.000 και επιχειρήσεις και όλο αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Όλες οι περιφέρειες έχουν ε, φορέα για την ανάπτυξή τους και είδα ας πούμε ένα παράδειγμα στην Κροατία όπου δημιουργήσαν ένα πρόγραμμα πιστοτικό για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Πώς τα κατάφεραν πήραν κάτι που είχαν χρησιμοποιήσει για κάτι διαφορετικό, διότι δεν μπορούσαν να αφήσουν όλες τις μικρομεσαίες να χρεοκοπήσουν, ή να, γιατί θα οδηγούσε σε μεγάλη ανεργία και βρήκανε λύση. Και αυτό σας δείχνει πόσο πολύ σημαντικές είναι οι περιφέρειες για την καταπολέμηση τη κρίσης. Ακόμη κάναμε μια άλλη ανασκόπηση προημερών για την ενέργεια και είχαμε ανταπόκριση από πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Σχεδόν όλες οι περιφέρειες, 90% σκέφτονται ότι η ενέργεια είναι ε, μεγάλη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Και βλέπουμε επίσης ότι οι παραλιακές περιφέρειες έχουν ήδη μεταβολή στο κλίμα και έχουν και σχέδια για την αντιμετώπιση τους. Η πράσινη ενέργεια, οι εναλλακτικέ ενέργειες, έχουν σημαντική θέση και δεν είναι μόνο θετικό αυτό για το περιβάλλον, αλλά όταν αποφασίζονται από περιφέρειες και ορισμένες περιφέρειες είναι πολύ δραστήριες, γίνονται πόλος ανάπτυξης για την περιφερειακή ανάπτυξη. Παραδείγματο χάρη, αν έχετε αυτοκίνητο βιομηχανία στην περιφέρειά σας, δημιουργείτε τις ανάλογες υποδομές που προσελκύουν και πολλούς άλλους. Έχουμε πολύ διαφορετικές λήξεις που διαπιστώνουμε, ανάλογα με τη γεωγραφική και φυσική, ε, τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιφερειών, που οπωσδήποτε παίζουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση και την καινοτομία. Μόλις γύρισα από το Belfort, που την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη γενική μας συνέλευση, ε, σε σχέση με την ενέργεια στην Ευρώπη, την απασχόληση, την καινοτομία κτλ. Τα συζητούσαμε όλα αυτά με ατέλειωτα παραδείγματα για τις ενέργειες των περιφερειών. Και, και η General Electric, ας πούμε, μια ε, πολυεθνική, ε, συμμετείχε, ήρθαν οι αρμόδιοι της Ευρώπης αυτής της εταιρείας να μας ζητήσουν τη συνεργασία μας και φτιάξαμε, οργανώσαμε με τη γενική μας συνέλευση στο εργοστάσιό τους. Και είναι πολύ σημαντικό που έχει αναγνωρίσει αυτή η πολυεθνική ότι στο περιφερειακό επίπεδο πολλές αποφάσεις λαμβάνονται για το ενεργειακό. 50 με 70% των προσαρμογών ε, γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, Σα τα πω όλα αυτά για να σας δείξω ότι οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αν έχουν τις σωστέ αρμοδιότητες. Σύντομα τώρα θα ήθελα να κάνω μια ακόμη ε, ε, παρατήρηση. Ε, κάναμε μια μελέτη για την αποκέντρωση και την οικονομική ανάπτυξη. Ήταν δύο ετών μελέτη, προσδιορίσαμε την αποκέντρωση, τους δείκτες για την αποκέντρωση, πολύ σημαντικό για μια μελέτη αυτού του τύπου και η χρήματοδοτική πόρη ήταν σημαντική. Κάναμε μία ανάλυση της Βασιλείας εάν η αποκέντρωση επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν στατιστικά σαφέστατα στοιχεία θετικής επίδρασης της αποκέντρωσης στην ανάπτυξη. Αν έχετε ένα συγκεντρωτικό κράτος, αυτό θα παρεμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτή είναι μια μελέτη που συζητήσαμε με πολλούς εμπειρογνώμενες, την υποβάλαμε και στην Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, τη συζητήσαμε με πολλούς ειδικού ε, της μακροοικονομικής και όλοι είχαν την ίδια άποψη ότι είναι πρώτη φορά που μια τέτοια μελέτη είχε γίνει και η μεθοδολογία ήταν απολύτως σωστά βασισμένη. Αξιόπιστη δηλαδή. Ένα ακόμη σχόλιο, ένα αποτέλεσμα ήταν ότι αναπτύσσονται καλύτερα οι περιφέρειες στην κοινοτομία όταν έχουν δυνατότητες έρευνας και πανεπιστήμια. Όταν όλα είναι συγκεντρωμένα σε μια χώρα, η καινοτομία και η έρευνα είναι πολύ πιο περιορισμένη παρά όταν είναι αποκεντρωμένη, διότι στο περιφερειακό επίπεδο ο ερευνητής συνεργάζεται με τις εταιρείες. Σας είπα λοιπόν διάφορα παραδείγματα των όσων πράττουμε και των ενεργειών μας. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Βεβαίως ασχολούμεθα και με την πολιτική συνοχής. Εδώ και πολλά χρόνια ξεκινήσαμε να ρωτάμε τα μέλη μας τι θα θέλανε. Ασχολούμεθα με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, Ξέρουμε δηλαδή πώς να τοποθετηθούμε για τη στρατηγική της Λισαβόνας και το μέλλον για το 2020. Επεξεργαζόμαστε τη μεταβολή του κλίματος, την ενέργεια, τις πληθυσμιακές μεταβολές, την χρηματοδότηση περιφαριακής ε, υγείας ε, στην Ανατολική Ευρώπη και στην ε, και στην Βόρεια Ευρώπη καταβάλλονται όλα από τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό. Δηλαδή η περιφέρεια καλύπτει 50% και πάνω στη Σουηδία φτάνουν στο 90%. Η χρηματοδότηση λοιπόν της ε, περιφερειακής δημόσιας υγείας οι ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες, η διαχείριση εκτάκτων αναγκών, η χρησιμοποίηση λιγότερων ε, γλωσσών, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η καινοτομία. Δεν μπορείτε μονίμως να εκπαιδεύετε μηχανικούς και ειδικού που ξέρουν πώς να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Ε, θέλετε βεβαίως ανθρώπους με σωστή κατάρτιση, επιχειρηματικότητα, πολιτική για την νεολαία, ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι τα χρόνια, έχουμε ε, δραστηριοποιηθεί σε πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα και στο τέλος του ε, περασμένου έτους δημιουργήσαμε μία ομπρέλα ενός δικτύου που είναι ένα δίκτυο νεολαίας ε, οι ενώσεις νεολαίας μπορούν να συμμετάσχουν συνεπώς στις εργασίες μας από καιρού εις καιρών όπως η πολιτική. Συνεργαζόμαστε για την αποκέντρωση με τη UNDP, ειδικότερα για τη μεταβολή του κλίματος και την ενέργεια. Πιστεύω άλλωστε ότι οι περιφέρειες στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσουν ένα ορόσημο ε, για περιφέρειες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη πολλά άλλα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίσαμε τι περιμένουμε από τη νέα Κομισιόν ε, για τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό κτλ. Ακόμη φροντίζουμε για τη διάδοση της επικουρικότητας στην Ευρώπη και την εφαρμογή της επικουρικότητας ενότητας στους πολίτες και στους θεσμούς με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για το κάθε θέμα που μόλις σας ανέφερα, τι κάνουμε. Έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από πολλές προσεγγίσεις. Μπορεί να οργανώσουμε και μια συνάντηση αλλά αναμειγνύουμε τις ε, ενέργειές μας και συμμετέχουν πολλά μέρη. Για το καθένα από αυτά τα θέματα λοιπόν δεν είναι ότι κάποια στιγμή καταλήγουμε σε μία τοποθέτηση ε, ή ότι οργανώνουμε μία διάσκεψη ή μία παρακολούθηση. Θέλουμε τα θέματα να γίνονται καλά κατανοητά από τις περιφέρειες και να εφαρμόζονται από τους επικεφαλείς των περιφερειών για την ανάπτυξη των πολιτικών τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Αυτά λοιπόν κάνουμε για τις περιφέρειες. Επαναλαμβάνω ότι οι περιφέρειες στηρίζουν η μία την άλλη. Ιδίως για την κατάρτιση, για την ε, δεν μιλάμε ε, για ειδικού, για εμπειρογνώμονες ή καθηγητές. Έχουμε ανταλλαγή μεταξύ των επικεφαλής, των ηθινόντων, των περιφερειών που έχουν συνηθίσει να εργάζονται μέσα σε μια διοίκηση με τους πολίτες κτλ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και με τη συνθήκη της Λισαβόνας ελπίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορέσει να κάνει περισσότερα πράγματα για να δώσει αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Ξέρω ότι έχει υπάρξει ε, μία προσπάθεια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, τις ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι ευκαιρία οι εκλεγμένοι των περιφερειών να γίνουν οι εταίροι σας. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία ανθίζει σε πάρα πολλές περιφέρειες, σε πόλεις και όχι μόνο σε συγκεκριμένους τόπους. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κλάους. Είχαμε προβλέψει μια ώρα από την συνεδρίασή μας για το θέμα αυτό, για να έχουμε και μισή ώρα περιθώριο για συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρον το ότι μας εξήγησε και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στις περιφέρειες δηλαδή. Ότι διανταποκρίνονται στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ήδη έχουν στήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι. Και παρακαλώ όποιος ενδιαφέρεται να γραφεί στον κατάλογο. Ο κύριος Μπλάσακ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και είμαστε υπεύθυνοι για τη συνεργασία αυτή από πλευρά. Είμαι υπεύθυνο μάλλον από την ε, Επιτροπή μα για τη συνεργασία αυτή. Ε, και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε συνεργασία σε επίπεδο Επιτροπή των Περιφερειών και με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, με το αντίστοιχο Συμβούλιο. Και δεύτερη ερώτηση, σημαντική συνεργασία, οι μηχανές και οι κινητήρες που αναπτύσσουν οι μηχανισμοί καλύτερα που αναπτύσσουν τα αστικά κέντρα. Κύριο Στρεμόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όντως ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος τη της Συνέλευσης των Περιφερειών. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που είναι επί της ουσίας των πολιτικών που καλούμαστε να προσαρμόσουμε και εμείς και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή τελευταία γίνεται μια συζήτηση και κάποιοι υποστηρίζουν την ε, επανεθνικοποίηση της πολιτικής ε, συνοχής. Σας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα και τι θέση έχετε. Thank you, Madame Благодаря. Я ще говоря на, български Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ε, ευχαριστήσω και εγώ, Πρόεδρε, για τις προτάσεις σας. Και θα ήθελα να ρωτήσω. Συγγνώμη, αλλά έχουμε πρόβλημα τεχνικό με τα μικρόφωνα. Δεν ακούγεται καλά η ομιλητρία. Θα δοκιμάσω λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα. Τώρα, τώρα είμαστε εντάξει, λέει πρόεδρος. για τη διαδίδωση αυτής της πληροφορίας στους εκπροσώπους της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης Είχατε μιλήσει λοιπόν για διάφορες πολιτικές Συγγνώμη που διακόπτουμε και πάλι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τα κανάλια της μετάφρασης. Μπερδεύονται τα διάφορα κανάλια μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχή λοιπόν που εφαρμόζεται. Είναι κομμάτι της δουλειάς σας στις περιφέρειες και θα ήθελα να μάθω εάν σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει στην αρχή της αλληλεγγύης στην πράξη και θα ήθελα να μάθω εάν προβλέπετε συγκεκριμένες δράσεις για τα νέα κράτη-μέλη. Είναι διαφορετικές μεταξύ τους περιφέρειες, έχουν σημαντικές αποκλίσεις να παρουσιάσουν μεταξύ τους. Προβλέπετε λοιπόν εσείς κάποια πολιτική ε, προσαρμοσμένη, προσανατολισμένη προς τις περιφέρειες των νέων κρατών μελών, ιδιαίτερα. Και ως προς τα κράτη, μέλη, εταίρος σας ποιος είναι, οι οργανώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, έχετε κάποια εταιρική σχέση μαζί τους. Και σκοπε... αν όχι σκοπεύετε να αναπτύξετε εταιρική σχέση με τις ε, με την τοπική αυτοδιοίκηση των νέων κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλώ τον Κλάους να απαντήσει, κύριο Κλίπ. Ναι, όχι μόνο συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε χωρίς αυτήν. Η πρώτη μας δραστηριότητα, σαν λόμπι αν θέλετε, ήταν η δημιουργία της Επιτροπής των Περιφερειών. Καθημερινή συνεργασία έχουμε. Το ίδιο και για το Συμβούλιο ή Κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τώρα, χάρη στην ε, Επιτροπή των Περιφερειών έχουμε νομίζω να ε, σημειώσουμε, μάλλον χάρη στη συνέλευση των περιφερειών έχουμε αυτή την πρόοδο συμμετέχουν και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Επιτροπή των Περιφερειών και το Συμβούλιο στην οργάνωσή μας. Όποιος επιλέγει είναι μέλος και αποστέλλεται πολιτικός ανάλογα με τη δραστηριότητα που αναλαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε και την επικοινωνία με τις περιφερειές μας. Γιατί οι άλλες διοργανώσεις που είναι συμβουλευτικά όργανα έχουν εκπροσώπους, μια μικρή ομάδα εκπροσώπων, που ε, εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές ενώσει, νομαρχίες, ε, διαμερίσματα ανάλογα με τη δομή της κάθε χώρας, αλλά είναι τελείως διαφορετική η εκπροσώπηση στο επίπεδο της, εκπροσώπησης. Εδώ έχουμε ένα δίκτυο συνεργασίας με τα αστικά κέντρα, με, τις... με τους δήμους. Βεβαίως είναι μέλη, περιφέρειες μέλη και οι δήμοι, όμως περισσότερο τώρα συνεργαζόμαστε μέσα του EuroCities, που είναι το δίκτυο των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της Ευρώπης επειδή μερικές φορές μπορεί να διαφωνούμε σε ορισμένα ζητήματα, πλην όμως καταρχήν τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε, στην ίδια κατεύθυνση βαζίζουμε. Και έχουμε αντιληφθεί και η δική του γραμματεία και εμείς ότι έχουμε κάθε συμφέρον να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Είναι κάτω αυτονόητο επομένω. Για τον κύριο Τρομόπουλο, επανεθνικοποίηση. Ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά είμαστε εναντίον της εναντίον τη πρόταση αυτή. Έχουμε απευθύνει μια ανοιχτή επιστολή πριν από δύο εβδομάδε περίπου στον κύριο Γκουμπαρόσο για το λεγόμενο non-paper, που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει, αλλά όλοι συζητούν. Και εν τέλει συζητήσαμε μαζί με άλλε ενώσει, όπω και τη Eurocities μεταξύ άλλων, για να διατυπώσουμε μια κοινή θέση, όπου είπαμε ότι δεν είναι καθόλου καλή λύση. Είναι αντίθετη, είναι αντιπαραγωγική και σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα που σα ανέφερα νωρίτερα, όπου αναφέρεται, αν δεν απατώ, με 16 φορέ η επικουρικότητα. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ τη Ευρώπη και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πιο σοβαρά. Και τώρα ξαφνικά έρχονται και μα λένε για υπερεθνικοποίηση. Δεν γίνεται. Ε, και σε σχέση με αυτά που σας ε, είπα και νωρίτερα, αν θέλετε να κοιτάξετε τη μελέτη για την επανεθνικοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη, πώς μπορούμε να μιλούμε για επανεθνικοποίηση της περιφερειακής πολιτικής αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη, γιατί ουσιαστικά επανερχόμαστε τότε στην αζέντα της Λισαβόνας το 2000, αν θυμάστε που θα έπρεπε υποτίθεται να έχουμε φτάσει μέχρι του χρόνου να είμαστε η πιο ανταγωνιστική οικονομία της Ευρώπης, του κόσμου. Κάτι το οποίο συμφώνησαν μεταξύ του κυβερνήσει και κάποιοι αξιωματούχοι των Βρυξελών, αλλά δεν μίλησε στο λαό. Δεν μίλησε στου πολίτε για να μπουν μέσα αυτή την πολιτική. Γι' αυτό είναι λάθο επιλογή η επανεθνικοποίηση. Γνωρίζω φυσικά ότι σε ορισμένε χώρε και ιδιαίτερα στι ανατολικέ χώρε τη Ευρώπη, στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, υπάρχουν πιο ε, κεντρικά οργανωμένε δομέ. Όμω, εμεί προβάλλουμε πάντα το επιχείρημα ότι πρέπει να αποδοθούν περισσότερε ε, εξουσίες της περιφέρειας για να είναι και πιο διαφανής η δράση τους. Ένα παράδειγμα μπορώ να σα δώσω από τη Γαλλία, από το Στρασβούργο, το οποίο χρηματοδοτείται απευθεία από την Ένωση από το, ως πιλωτικό πρόγραμμα με 100% χρηματοδότηση απευθεία, ενώ οι υπόλοιπε περιφέρειε ε, χρηματοδοτούνται έμεσα από το κεντρικό κράτο δηλαδή, αλλά τελικά τα χρήματα πάνε πάλι πίσω διότι δεν απορροφούνται όπω πρέπει. Και μετά η κυρία Ισμίνοβα. Για την συνοχή δεν υπάρχει αμφιβολία φυσικά ότι δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών, να εργαστούμε για την αλληλεγγύη και φυσικά υποστηρίζουμε την πολιτική της συνοχής για τις πιο φτωχές περιφέρειες και ιδιαίτερα για τις πιο αδύναμες περιφέρειες. Υπάρχουν ε, προβλήματα ουσιαστικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ανταγωνιστικότητα βεβαίω, ναι, αλλά εμείς ζητούμε μια πολιτική τη συνοχής η οποία σημαίνει να σταθούμε στο πλευρό να προσφέρουμε αρρωγή στις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης και κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Μέλη μας είναι περιφερειακέ, δηλαδή δεύτερου και τρίτου επίπεδου εκπροσώπηση, περιφερειακές αρχές και μετά ανάλογα, αν χρειαστεί, μπορούμε να απευθυνθούμε και στην εθνική κυβέρνηση. Ελπίζω να πάτε στην ερώτησή σα. Ευχαριστώ πολύ, Λομπέρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη είναι η εξής. Μιλήσατε με ενθουσιασμό για την ενέργεια, το κλίμα κτλ. Αλλά αν εξετάσουμε μεγαλύτερη προσοχή αυτό το οποίο ε, αποτελεί κείμενο δαπάνης από τα περιφερειακά τα ε, χρήματα. Από το 2000 στο 2006 ήταν 2-3%, τώρα είναι 14%. Ε, Μόλις. Και το συνδυάζω με την έκθεση Μπάλκα που μιλούσε για το γεγονό πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα από τη βάση του, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και σε τελευταία ανάλυση μιλούσε ε, για τμηματοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ευρύτερα κονδύλια για συγκεκριμένους στόχους. Πω αυτά όμως μπορεί να είναι απολύτω αρνητικά από τη σκοπιά της ολοκληρωμένης προσέγγισης και του Περιφερειακού Ταμείου, για παράδειγμα. Ρωτώ, τι πιστεύετε, δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα χρηματοπιστωτικά μας ε, μέσα έτσι ώστε ε, να έχουμε πιο στοχευμένα κονδύλια, να έρχονται περιφέρειες και να ψωνίζουν αν θέλετε στις Βρυξέλλες ή να έχουμε μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση. Και δεύτερον, ε, είστε εδώ σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας προσκάλεσε, που προσκαλεί η Προεδρία της οργανώσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικές. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δική μας ατζέντα. Με ποια έννοια. Τις εκθέσεις μας που είναι ζωτική σημασία για το μέλλον από άψη συνοχής. Μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτές τις εκθέσεις. Ξέρετε ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας μας. Ευχαριστώ. Κύριε Σπίπεν. Uh, Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω και εγώ σε αυτήν την ερώτηση. Ακούσαμε το τι πράττει η συνέλευση των περιφερειών. Αλλά εδώ έχουμε περισσότερο να συστήσουμε και τις σχέσεις ε, ως προς την νομοθεσία ε, και την, ε, με, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι το καινούριο προσφέρει δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας. Προς το συμφέρον φυσικά των περιφερειών της Ευρώπης. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Από εμάς τι περιμένετε. Συγκεκριμένα από την Επιτροπή μας. Τι προσδοκίες έχετε. Τους προσεχείς μήνες τι περιμένετε από εμάς. Θα ήθελα να ακούσω τι περιμένετε, όπως είπα. Δεύτερη ερώτηση. Εκθέση Μπάλκο. και τα όσα προεξαγγέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε, δείχνουν ότι ε, περισσότερο στο δημογραφικό, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό ε, ζήτημα θα στραφεί η περιφερειακή πολιτική. Οι υποδομές όμως, η ανταγωνιστικότητα, τι, που, τι γίνονται. Ευχαριστώ κύριος Ολένιτσακ. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να υποβάλω. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την αποκέντρωση, συμφωνώ απόλυτα αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, υπάρχουν ορισμένες, ε, ε, ορισμένα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Μιλήσατε για προσδοκίες και είπατε ταυτόχρονα ότι πρέπει να δυναμωθούν περισσότερο οι ε, περιφέρειες. Ναι, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των περιφερειών. Στα κράτη-μέλη βεβαίως. Αλλά αυτό σχετίζεται και με το ποιε είναι οι προσδοκίε και τι εννοείται συγκεκριμένα. τι, ε, πρέπει να πάρουν οι περιφέρειες ε, από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, πώς βλέπετε την πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε μία ε, στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα. Και έχω να κάνω εξή ερώτηση. Πώς πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η πολιτική προς τις μακροπεριφέρειες και ποια είναι η δική σας στάση απέναντι σε όλα αυτά. Uh, Ίσως θα μπορούσα να απαντήσω πρώτα απ' όλα στον κύριο Πίπερ. Και σας το συγγνώμη που μιλώ αγγλικά. Ε, που... Ναι, ε, ε μας ρώτησε ε, τι προσδοκούμε εμείς από εσάς, τι θέλουμε από εσάς. Ναι, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, για τη μελλοντική κοινωνική συνοχή, πολιτική συνοχής. Θέλουμε να σας δώσουμε την άποψή μας, άποψη που προέρχεται από την ε, λεπτομερή συζήτηση με τα μέλη για το μέλλον, ε, συνεργασία για το 2020, Λισαβόνα κτλ. Για τον προπολογισμό, το μελλοντικό προπολογισμό, για αυτό το ανεπίσημο έγγραφο, το non-paper που είδαμε, για μας ήταν σοκ. Κοιτάξτε, αν το διαβάσετε, πραγματικά μπορεί να πάθει καρδιακή προσβολή. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, αγωνιστούμε κατά αυτής της ε, ε, τοποθέτησης και νομίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε εταίροι εσείς και εμείς. Και δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για το περιβάλλον και την ατζέντα του Κέντενμπορ και τα λοιπά και μετά να ξεχνάμε τελείως την ανταγωνιστικότητα. Τώρα, όσον αφορά μια ερώτηση από τον Λάμπερ για τα χρήματα τα οποία δεν δαπανώνται. Ναι, αυτό είδαμε και στην έρευνα που στείλαμε στα μέλη μας. Είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι περιφέρειες δεν έχουν ε, χρησιμοποιήσει και εξαντλήσει πιθανές, ε, τα πιθανά κονδύλια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενεργειακή πολιτική, για παράδειγμα. Γιατί? Όχι ότι δεν εργάζονται προς την κατεύθυνση ενέργειας, ε, αντίθετα, είδαμε ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριε, αλλά δεν έχουν απαραίτητη πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά και διαφορετικά προγράμματα τα οποία τα χειρίζονται ε, διαφορετικές γενικές διευθύνσει και σύμφωνα με άλλε τόσε κατευθυντήριε γραμμέ, καταλαβαίνετε ότι μία ε, περιφέρεια πρέπει να γνωρίζει να, να τα βγάλει πέρα μέσα αυτή τη ζούγκλα των δυνατοτήτων επιδότηση. και αυτό είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αν η περιφέρεια είναι μεγάλη στο τέλο ε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι περιφέρειες και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επενδύουν και δεν εργάζονται το τομέα τη ενέργεια. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι υπάρχουν περισσότερε ισχυρέ και λιγότερε ισχυρέ περιφέρειες και για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι κομιτείε δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρέ, ε, ακολουθούν μια ενεργειακή πολιτική για τις δικές τους, ε, για τις δικές τους και στους πολιτικές ε, ε, και για τις κατοικίες τους, καταρτίζουν τους ανθρώπους, τα, τα παιδιά κτλ. Να καταλάβουν την ενέργεια, έχουν πράσινες ε, κρατικές προμήθειες. Προσπαθούν με δύο λόγια να εργαστούν με έναν τρόπο που να είναι αηφόρος, εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Δεν έχουν οι, οι, ε, οι ίδιες πόρους και όμως, από την άλλη, αν δείτε μια περιφέρεια όπως η Βαλένθια για παράδειγμα, που ε, ε, εκεί ήδη υπάρχει μια επένδυση ενός δις ευρώ για αιωλικά πάρκα, τα οποία ξέρουν πού θα τοποθετηθούν, πού θα κατασκευαστούν. Και έχουμε και πολλές άλλες περιφέρειες που έχουν προγράμματα επιδοτήσεων, ε, δίνουν φθηνότερες, φθηνότερα δάνεια σε ιδιώτες επιχειρήσεις για να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε, να χρησιμοποιήσουν καθαρές μορφές ενέργειας. Και κατά βάλλον θα προσπαθούν λοιπόν ξέρετε με το αν έχουν τα χρήματα ή όχι. Τώρα όσον αφορά την μακροοικονομική προσέγγιση που επίσης αναφέρεται στο ανεπίσημο έγγραφο. Εδώ πραγματικά είναι τελείως λάθος να προβλέψουμε μεγάλο κοντήλια, γραμμούμε το Α για αυτό το θέμα, το Β για το άλλο. Το θέμα δεν είναι η διανομή χρημάτων. Είναι ε, διαφορετική αντιμετώπιση και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είστε ε, διευθυντής μιας επιχείρησης και θέλετε να πουλήσετε ε, αυτοκίνητα αξία 50 δις ευρώ. Μα άμα δεν έχετε πολιτές δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, να ξέρετε τις προθέσεις σας. Και εδώ ε, καταλαβαίνετε πρέπει να δούμε τους δικούς μας πολιτές. Ε, δεν μιλάω μόνο για περιφερειακούς πολιτικούς, ε, που βεβαίως εμπλέκονται, αλλά το να δώσουμε τα, αυτά τα μεγάλα ποσά κάπου και να πούμε ε, τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο του, λυπάμαι, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Πρέπει να σκεφτούμε και ποιοι θα υλοποιήσουν τι πολιτικέ. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που θέλετε. Και για να, όσον αφορά την αλλαγή τη ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι, δεν το πιστεύω. Το ερώτημα είναι. Ε, το ερώτημά σας είναι αν παρακολουθούμε την εργασία σα. βεβαίω παρακολουθούμε το τι κάνετε. Αλίμονο, με ιδιαίτερη προσοχή. Και εδώ και μια άλλη ερώτηση από εδώ, ναι, από Ναι. Ποιε θα είναι οι πλέον αρμοδιότητε που θέλουμε να, να πάρουν οι περιφέρειε. Πολύ λεπτό θέμα βεβαίω. Επικουρικότητα, αποκέντρωση, διαφοροποίηση. Δεν τολμάμε να πούμε στα μέλη μα ε, οργανώστε τι περιφέρειες στη χώρα σα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να το υπαγορεύσουμε αυτό. Αλλά εάν ε, κοιτάξετε τι υφιστάμενε μελέτε, όχι μόνο τι δικέ μα, αλλά και του ΩΣΑ, που δείχνουν ότι οι περιφέρειες ε, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη οικονομία. Αν εξετάσετε λοιπόν τέτοια θέματα, αν εξετάσετε το πώς θα εφαρμοστεί η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε που θα προκύψουν τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες οι περιφέρειες. Κατά την άποψή μου, αρμοδιότητες αυτές πρέπει να είναι πολλές. Και τέλος, όσον αφορά την στάση μας προς την πολιτική για τις ε, πιο ε, απομακρυσμένες περιφέρειες, τις μακροπεριφέρειες, ναι, το συζητήσαμε από μακρόν, λέει και η Πρόεδρος. Προσπαθούμε να ε, έχουμε ερετούς πολιτικούς της περιφέρειας που να λαμβάνουν τις πραγματικές αποφάσεις που θα αλλάζουν ε, την καθημερινή ζωή. Και εδώ δημιουργούμε τις, ε, αυτές τις, αυτούς τους φορείς της τις που έρχονται και όλοι μαζί και συμφωνούν και μη την βαλτική περιοχή θα δείτε ότι όλα αυτά είναι ωραία. Τα συζήτησαν και στο γραφείο μας πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν και πολλοί σκανδιναβοί πολιτικοί δεν είχαν ακούσει ποτέ για αυτό το ζήτημα. Μα αυτό είναι διαβούλευση με του περιφερειακού πολιτικού, δεν το πιστεύω. Και όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε η διαβούλευση, αλλά κοιτάξτε, πάρτε την απόφαση από τα χέρια των αιρετών πολιτικών, βάλτε το, δώστε την απόφαση σε κάποιους φορείς και θα χαθείτε όλοι. Κανείς δεν θα ξέρει ποιος αποφασίζει γιατί. Και αν εσείς ως πολίτες δεν ξέρετε πλέον ποιος είναι υπεύθυνο, το μόνο που αισθάνεστε είναι θυμό και κάποια στιγμή θα πείτε δεν με νοιάζει, α κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ έτσι κι αλλιώ ε, ε, δεν πρόκειται να με ακούσουν. Αλλά εάν δεν, ε, ε, δεν καθαρίζονται οι δρόμοι σωστά στην περιοχή σα, ξέρετε ποιο θα πάρετε τηλέφωνο. Αν όμω πρόκειται για κάποιον ανώνυμο φορέα που τα έχετε αναλάβει όλα αυτά, τότε αισθάνεστε και εσείς ανήμπορος και δεν κάνετε τίποτα και καταλαβαίνετε πού θα βρεθούμε. Γι' αυτό έχουμε ένα πρόβλημα με αυτές τι μακροπεριφέρειε. Και κάτι άλλο. Αν ξεκινήσετε μια στρατηγική προ την κατεύθυνση αυτή, να τη σκεφτείτε μέχρι το τέλο. Γιατί έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 μελών. Θέλετε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 10 τέτοιων φορέων στο μέλλον, 10 μακροπεριφερειών. Αυτό, αυτός θα είναι ο στόχο μα. Και βεβαίω δεν είναι μακροπεριφέρειες και μακροχώρε. Δεν μου αρέσει η λέξη μάκρο ε, περιφέρεια. Μιλάμε για συνεργασία με τις ε, κυβερνήσεις. Έχουμε την Βαλτική, το Δούναβι ε, και τι άλλε περιοχές και μετά δεν βρισκόμαστε πλέον όλοι μαζί. Ε, και φτιάχνουμε έτσι αυτές τις μακροομάδες. Λοιπόν, τι να σας πω. Ε, και βασίλευε τελικά. Αυτό θέλουμε όλοι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μικαλτόιρεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που θέλω να σας υποβάλω. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δημιουργήσει ένα φορέα που είναι υπεύθυνο για την ε, εδαφική συνεργασία. Αυτό ήθελαν οι περιφέρειες. Ήθελαν ε, την οργάνωση σε διασυνοριακό επίπεδο προς την κατεύθυνση ανάπτυξης η δική σας η οργάνωση πώς βλέπετε αυτές τις προσπάθειες. Πιστεύετε ότι αρκούν ή χρειάζονται να κάνουμε κάτι άλλο. Και επίση εσείς συζητάτε το θέμα της συνοριακής συνεργασίας. Όταν τα σύνορα είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα. Γιατί εδώ μιλάμε για νομοθεσία άλλων χωρών. Επόμενος ομιλητής, κύριος Μπλάντμπερν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω μια ερώτηση και δεν θέλω να κάνω σχόλια, αν μου επιτρέπετε, σε αυτά τα οποία είπε ο μιλητή μα. Είπε ότι η συνέλευση ασχολήθηκε με το δεύτερο σκέλος. Αλλά εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε σε αποκεντρωμένα κοινοβούλια, Σκοτία και Ιρλανδία, αλλά τα υπόλοιπα στηρίζονται στις τοπικές κυβερνήσεις. Εσείς δηλαδή, να ρωτήσω το εξή, αναγνωρίζετε τις τοπικές αρχές, ως ισοδύναμες αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και ένα σχόλιο τα. Και χαίρομαι γιατί σε απάντηση σε μια προηγούμενη ερώτηση είπατε ότι δεν θέλετε να δώσετε σε αρμοδιότητε στι περιφέρειε. Και να σα πω κάτι, το κόμμα μου ε, θέλει να καταργηθούν τελείω οι περιφέρειε ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και να δοθούν πάλι εξουσίε και αρμοδιότητε στι τοπικέ αρχέ. Γιατί οι περιφέρειε δεν ήταν καθόλου αποδοτικέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν γιατί δεν προχωρήσετε περαιτέρω το ζήτημα για περισσότερη αποκέντρωση ισόφελα των περιφερειών. Γιατί κάτι τέτοιο θα με δυσαρεστούσε ιδιαίτερα, σα το λέω. Τώρα, ένα άλλο σχόλιο που έχω να κάνω και θα είμαι σύντομο είναι το εξή. Ε, το θέμα τη περιφερειακή πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα τη χρηματοδότηση. Είναι κάτι που και εσεί το εντοπίσατε όταν ε, μιλήσατε για τα πειράματα και τα πιλωτικά σχέδια Αναφερθήκατε στην περιοχή του Στρασβούργου, νομίζω, όπου η ίδια περιφέρεια τη Αλσατία δαπανά τα χρήματα και τα παίρνει απευθεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μάθω το πώ ε, όλα αυτά ε, ε, εφαρμόζονται ως έννοιε σε επίπεδο τοπικής, ε, τοπικών αρχών. Γιατί εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε φορείς που ασχολούνται με την περιφερειακή χρηματοδότηση και που στην ουσία τα, κάνουν θάλασσα σε γενικέ γραμμέ και δημιουργούν τρομερά προβλήματα ε, στι τοπικέ αρχέ με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα σχέδια. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα ήθελα να μάθω και τη δική σα άποψη. Ποιο πιστεύετε θα ήταν ο πιο κατάλληλο τρόπο για να προχωρήσουμε προ τα μπρο, δεδομένου του γεγονότο ότι δεν έχουμε επανεθνικοποίηση. Δεν είμαι σίγουρο κατά πώ θα γίνει κάτι τέτοιο, πάντω ανεξάρτητα με τι θα γίνει, θα υπάρξει διαθέσιμη χρηματοδότηση στα επιμέρου κράτη-μέλη. Και σίγουρα θα ήθελα να μάθω πώς βλέπετε αυτό το είδος της χρηματοδότησης ε, και αν βλέπετε να αποτελεί αντικείμενο διαχείριση σε πολύ τοπικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Κόρτες Λάστρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Στον εκπρόσωπο της ε, Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, δυνατότητα διακυβέρνηση, ε, ποια εργασία πραγματοποιείται προ την κατεύθυνση αυτή για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, μα απασχολεί ιδιαίτερα. Δεύτερον, ποια είναι η άμεση σχέση σα με την κοινωνία των πολιτών. Καταλαβαίνετε, πώ έρχεστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Um... Ευχαριστώ όσον αφορά το ETTC. Είναι το Ινστιτούτο Νομικό Ινστιτούτο για την Εδαφικότητα. Είναι, κάτι το οποίο έχουμε προαθήσει εξ αρχής ουσιαστικά με τον Γιάνν Ουρμπριθ που ήταν εισηγητής εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε οργανώσει την τότε ακρόαση. Με άλλα λόγια είμαστε υπέρ αυτού του φορέα. Βεβαίως χρειάστηκε χρόνος να προσαρμοστεί με την πραγματικότητα, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά γύρω από τα Πυρηναία τώρα ε, προχωράνε μεταξύ των περιφερειών που ε, χαρακτηρίζονται από παρόμοια γεωγραφικά χαρακτηριστικά και άλλα χαρακτηριστικά και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Είμαστε υπέρ λοιπόν Τώρα, κατά πόσο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στο πλαίσιο του Euro District, ενδεχομένως ναι, αλλά δεν έχουμε άποψη γιατί θέλουμε να δούμε περισσότερα παραδείγματα αφού λειτουργήσει το σύστημα το προηγούμενο. Όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, θα ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι ξέρετε ότι στον κανονισμό υπάρχει ε, υπάρχει πρόβλεψη ότι όσες χώρες είναι εκτός ΕΕ μπορούν να συνάψουν συμφωνία με την ΕΕ για να συμμετέχουν οι περιφέρειές τους. Αυτό το θέλαμε εξ αρχής γιατί θέλαμε να μείνουμε ανοιχτοί σε μέλη εκτός ΕΕ. Τώρα, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλη αυτή η συζήτηση ομολογώ και ίσως καλύτερα να πιούμε μια μπύρα μαζί και να το συζητήσουμε διότι έχετε δίκιο Έχετε το ε, σκοτσέζικο εκτελεστικό, τη Βουλή. Εμείς δεν έχουμε το σκοτσέζικο εκτελεστικό, ούτε τη Βόρεια Ιρλανδία. Τώρα, αν ε, ρωτήσω τα μέλη μου, μπορείτε να μου εξηγήσετε το Ηνωμένο Βασίλειο, η νομοσπονδία, η νομοσπονδία, τι είναι νομικά, κανένας δεν θα ξέρει. Ε, απλώς την πραγματικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου γνωρίζουμε είμαστε υπέρ της εκχώρησης περισσότερων εξουσιών στην περιφέρεια. Η περιφερειακή αρχή είναι το δεύτερο επίπεδο εκλεγμένων αρχών στις περισσότερες χώρες και ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάτι τελείως, διαφορετικά, τελείως διαφορετικό, ένα γραφειοκρατικό σύστημα ανώνυμο που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνο γιατί διαχείριση κονδυλίων. Το παράδειγμα που σας έδωσα ήταν η περιοχή της Αλζάς στη Γαλλία. Δεν είναι ε, το μόνο παράδειγμα, αλλά σε πολλές χώρες ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες. Καμιά φορά υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι πάντα χάλια τα πράγματα της διαχείρισης, αλλά ε, κοιτάξτε τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Είναι πολύ χειρότερες καμιά φορά. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, προτιμώ να έχετε 10 διαφορετικούς ανθρώπους ε, στις περιφέρειες να ασχολούνται με τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και να έχετε δύο προβληματικές περιφέρειες και να μην ε, έχετε μία κυβέρνηση η οποία τα πάει χάλια <coughs> και οι συνέπειε είναι για τον ολόκληρο το λαό. Έτσι είναι η ζωή. Λάθη υπάρχουν πάντοτε. Όσον αφορά τώρα τη διακυβέρνηση, τη συνέλευση, μιλήσαμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, γιατί είναι σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι αυτό απαντά και στην ερώτηση. Ε, θέλουμε πραγματικά να έχουμε συνεργασία μεταξύ εθνικής κυβέρνησης, ευρωπαϊκών φορέων και περιφερειών. Τώρα, η κοινωνία των πολιτών. Καλή παρατήρηση, ενδιαφέρουσα παρατήρηση με την έννοια ότι όσα συμβαίνουν σήμερα στο επίπεδο των περιφερειών στην Ευρώπη βλέπουμε ότι οι πολιτικοί των περιφερειών λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχουμε πολιτικές ομάδες, ούτε εθνικέ ομάδες. Πολύ συχνά έχουμε πολύ ανοιχτέ συζητήσεις μεταξύ πολιτικών και εκλεγμένων και βλέπετε ότι οι πολιτικοί από το ίδιο κόμμα σε μια χώρα έχουν τελείω διαφορετική άποψη. Είναι ρεαλιστικές πλέον οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ στελεχών και εκλεγμένων. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία είναι πολύ σημαντικό στην, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, ε, χρειαζόμαστε να συνεργαστούμε περισσότερο με το ΕΚΟΣΟΚ. Ε, πολύ συχνά καλούμε στις δραστηριότητες της συνέλευσής μας, αν πρόκειται για ενέργεια, νεολαία κτλ. Καλούμε, λέω, ε, πρωταγωνιστές της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν, διότι υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ των όσων πράττουν και του περιφερειακού επίπεδου. Είναι θαυμάσια παραδείγματα όσον αφορά την εφεύρεση λύσεων για κάθε τύπο ε, περιφερειακών προβλημάτων όπου η κοινωνία των πολιτών συνεισφέρει με πολύ ενδιαφέροντο τρόπο. Τώρα, οι δυνάμεις των πολιτών είναι ένα άλλο θέμα ε, είναι οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συζητάνε μεταξύ τους. Έχω πρόβλημα, λέει η Πρόεδρος. Έχω ακόμη έξι συναδέλφους που θέλουν ε, το λόγο. Ήδη έχουμε πάρει χρόνο από το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συνοψίσουμε λοιπόν τα σημερινά και τα αυριανά θέματα στην ημερήσια διάταξη μάλλον θα τα συντομεύσουμε για να μπορέσω να δώσω το λόγο στους έξι συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ όμως να είστε πάρα πολύ σύντομοι και εσείς και ο επισκέπτης μας στις απαντήσεις του. Ο κύριος Μποστινάρο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την τοποθέτησή σας όσον αφορά το μη έγγραφο της Κομισιόν. Πρώτη ερώτηση. Τι, ποια είναι η προσέγγιση σας για την πολιτική συνοχής. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές σας. Δεύτερον, είστε έτοιμος τώρα να συνεργαστείτε στενά με την ομάδα εργασίας για την πολιτική συνοχή στη μελλοντική που θα συστήσουμε στην Επιτροπή μας. Άλλη ερώτηση τι επιπτώσεις πρέπει να έχει η πολιτική συνοχή μέσα στο νέο νομικό πλαίσιο εν ώψη των δημοσιονομικών περιορισμών. Τι έχουμε και οικονομική κρίση και το μέλλον του πλαισίου του οικονομικού ε, είναι αυτό που είναι. Τέλος. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πρόθυμος να γεφυρώσουμε ότι χάσμα υπάρχει με την περιφερειακή διάσταση, διότι η διάσταση αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει διαπεριφερειακό συντονισμό και ενδοπεριφερειακό συντονισμό. Δηλαδή χωρίς την περιφερειακή διάσταση τίποτα δεν προχωράει. Ο κύριος Μάιερ και μετά ο κύριος Γκούλμαντς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ στο δυνατόν σύντομο. Καταρχά, ω Αυστριακό, θα πρέπει να ρωτήσω το Γενικό Γραμματέα και εγώ εάν υπάρχουν επαφέ με τον μελλοντικό επίτροπο, τον κύριο Χάνεν, και αν έχει κάτι να μα δώσει από το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τι προσδοκίε ε, που έχετε από τον νέο επίτροπο, από τη δουλειά του νέου επιτρόπου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μια οδυνηρή ερώτηση. Αν κοιτάξετε τα χρήματα, τα κονδύλια, τα κονδύλια για τη συνεργασία είναι μόνο 2% από όλο το, τα κονδύλια της συνοχής. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. 2%. 2,20 για την ακρίβεια. 7,7 δις για το 2007-2013. Αν πάρετε την προηγούμενη πρόπτικη θα βλέπατε ότι η εδαφική συνεργασία στην οποία συμμετείχαν πολλές χώρες δεν ε, υλοποιήθηκε σε 95% αλλά στο 91%. Δηλαδή κατά 4% δεν υλοποιήθηκε. Καλύτερα σε άλλες κάποιες χώρες αλλά χειρότερα και σε κάποιες άλλες. Δεν υπάρχουν, ε, υπάρχουν στοιχεία για τη νέα προοπτική αλλά η βελτίωση του συστήματος διοικητικού ελέγχου για τα εδαφικά σχέδια από 105 μη απορριφθέντα ε, σχέδια, τα 25, είναι εδαφικά. Δηλαδή, η ερώτησή μου τελικά είναι η εξής. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε εσείς και εμείς για να βελτιώσουμε αυτό το πράγμα. Είναι 2% των κονδυλίων, αλλά πολύ ευαίσθητα κονδύλια, γιατί πολλές χώρες συμμετέχουν σε αυτά τα σχέδια και μοιάζουν τα, τα σχέδια συνοχής, τα εθνικά, να μένουν πίσω και τα κοινωνικά συνοχής και τα λοιπά. Ε, συμφωνείτε με την ανάλυση μου βάσει των στοιχείων που έχετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Η μελλοντική μας πολιτική συνοχής. Έχουμε μία τοποθέτηση την οποία εγκρίναμε. Α, εσείς μου ε, με ρωτήσατε, ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα σχετικό έγγραφο, δεν θα στο διαβάσω. Αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο κτλ. κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα στη συνέλευση και το αναπτύσσουμε περαιτέρω. Πράγματι, θέλουμε να συνεργαστούμε όσο πιο στενά γίνεται μαζί σας δημοσιονομικοί περιορισμοί. Ναι, υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι μια πολύ σημαντική συμβολή για να βγούμε από την κρίση είναι το γεγονός ότι οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν την προσωπική τους πολιτική ανάπτυξης. Βεβαίως, από πού προέρχεται η οικονομική ανάπτυξη, ποιος πρόχνει για καινοτομία, είδαμε από την ανασκόπηση σε σχέση με την οικονομική κρίση ότι οι εταιρείε που ήταν πολύ καινοτόμε, που πέρασαν από μεγάλε μεταβολές για να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό κτλ. Οι εταιρείε αυτές επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Ο νέο επίτροπο. ναι. Το άκουσα την Παρασκευή στη μέση μια συνέντευξη τύπου και σχεδόν αναπήδησα, διότι η νέα Επίτροπης, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής προέρχεται από περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε όλες τις περιφέρειες από την Αυστρία σαν μέλη και επεξεργαζόμαστε την επικοινωνία μαζί του προσδοκίες τώρα πολλές έχουμε, περισσότερες προσδοκίες από όσες μπορεί να εκπληρώσει ο Επίτροπος. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πολιτική της Τανούτα Χούπνερ, η οποία έκανε θαυμάσια εργασία πιέζοντας για τις περιοχές, περιφέρειες, με Όσον αφορά την εδαφική συνεργασία και την διαπεριφερειακή, ε, όσα είπατε δεν είναι αληθή, μικρό ποσό, μικρά κονδύλια, περισσότερο ίσως στο μέλλον, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και την προσέγγιση. Δηλαδή στην Ευρώπη μιλάμε πάντοτε για την ποικιλομορφία, τον πλούτο, των πολιτισμών μας και ε, τη σημαντική συμβολή του για το μέλλον, αλλά στο τέλος όταν θέλουμε να συνενώσουμε τους ανθρώπους και να λειτουργήσουν μαζί έχουμε πρόβλημα. Και το τα εδαφικά σχέδια είναι θαυμάσια για να προχωρήσουμε προς αυτή την ε, ε, κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει να κάνουμε ανταλλαγή εμπειριών. Θα έπρεπε να έχουμε σχέδια με την συμμετοχή περιφερειών από περισσότερες χώρες για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος και τα κονδύλια που δίνονται γι' αυτό είναι σχεδόν, σχετικά περιορισμένα. Γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώξουμε μελλοντικά. Στις συζητήσεις που έχουμε και στις συναντήσεις μεταξύ πολιτικών, άσχετα με τα πολιτικά κόμματα από τα οποία προέρχονται, είναι καλοπροετοιμασμένοι, ξέρουν τις πολιτικές τους στο κράτος τους και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από συναδέλφους από άλλες χώρες και αναρωτιούνται από πού ξεπηδάνουν αυτές οι διαφορές. Προσπαθούν λοιπόν να καταλάβουν το όλο ιστορικό και αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν προέρχεται από διαφορετική χώρα και διαφορετικό περιβάλλον υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικές πραγματικότητες οι οποίες επηρεάζουν και στη συζήτηση τελικά διαπιστώνεται ότι ε, επιτυγχάνεται υψηλότερη ενημέρωση γιατί προσλαμβάνεται περισσότερες πτυχές. Και νομίζω ότι η εδαφική συνεργασία ακριβώς θα μπορούσε να παράσχει καλύτερες λύσεις περιφερειακές. Ε, και είναι μια επίκριση και προς τον φορέα μας. Αυτή η πολιτική υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Πάντοτε έχουμε κάποιο φυλάδιο, κάτι στο διαδίκτυο και έχουμε, αλλά αυτοί που συμμετείχαν δεν μπόρεσαν πραγματικά να αφομοιώσουν τις καλύτερες και πιο πρόσφατες γνώσεις και να τις επικοινωνήσουν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προ, το, προχωρήσουμε. Ο κύριος Λούχαν, τελευταίος ομιλητής. Θα ήθελα μια ερώτηση σε σχέση με το ε, ΑΕΠ το οποίο διαρκώς καταραίει σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε λοιπόν ότι μειώνεται διαρκώς το ΑΕΠ και ως εκ τούτου θα μειωθεί και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή όμως η Επιτροπή συζητά άλλες προτεραιότητες. Την περιβαλλοντική ρήπανση, τη δημοσιονομική κρίση, το περιβάλλον, την ε, ύπεθρο. Ε, σε ποιο βαθμό λοιπόν θεωρείτε εσείς ότι αυτή η πτυχή μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις της περιφέρειας και δεύτερον και την περιφερειακή ανάπτυξη πάνω απ' όλα και δεύτερον εσείς συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε η περιφερειακή ανάπτυξη να εξασφαλίσει τα κονδύλια για τον στόχο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Σας ευχαριστώ. Thank you, Madame Σας ευχαριστώ. Αν θέλει να απαντήσει, ε, αν θέλει η τελευταία ομιλήτρια να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα νέα προγράμματα σας στόχο έχουν η κυρία Λουκασίετσκα ε, κολάρσκα, συγγνώμη, έχουν σαν στόχο να ε, περιορίσουν τις αποκλήσεις μεταξύ των περιφερειών. Είναι σχεδιασμένα μερικά από αυτά, ειδικά για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των περιφερειών. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα ειδικά για την Ανατολική Ευρώπη με τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Και θα ήθελα να και συζητούμε την ε, μελλοντική περιφερειακή πολιτική, να δω τι είδου συζήτηση θα αναπτυχθεί για τέτοιου είδους μέσα Εσείς είστε σε θέση να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους προγραμμάτων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, παράδειγμα, που ονομάζεται Πρόγραμμα για την Ανατολική Ευρώπη. Κάποια κονδύλια για συγκεκριμένα και συγκεκριμένες δύο περιφέρειες. Μιλάτε για την, για την ανατολική εταιρική σχέση. Όχι, είναι η απάντηση. Μιλάω για ένα ειδικό περιφερειακό πρόγραμμα έκτακτο και ιδιαίτερο σχεδιασμένο για τις περιφέρειες αυτές. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια ιδέα για την αποτελεσματικότητά του. Η κυρία Μουκατσίρσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μίλησατε για την Ευρώπη των πολιτών, για την αποκέντρωση, την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, Ο δικαιούχος όμως για να αξιοποιήσει τα κονδύλια θα πρέπει να έχει και πρόσβαση σε αυτά. Όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ περίπλοκες διαδικασίες, γραφειοκρατικές, και ερωτώ τι είδου μέτρα λαμβάνετε ή μπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε τη γραφειοκρατία, να καταστήσετε πιο απλή την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί εγώ πολύ συχνά αντιμετώπισα στο παρελθόν ανόητες διαδικασίες και κανονισμούς ή διατάξεις καλύτερα οι οποίες παρεμποδίζουν οποιονδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση στα κονδύλια ή καθιστούν την κατάσταση πολύ δύσκολη. Τα δε προγράμματα για τη βελτίωση της, ε, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρήπανση ή αντίστοιχα άλλα τέτοια περιβαλλοντικά προγράμματα θα πρέπει να αποτελούν όχι βάρος αλλά κέρδος για τις περιφέρειες όπως το Natura 2000 όπου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τις περιφερειακές αρχές να έχουν πρόσβαση στο Natura 2000 και στα κονδύλια του. πριν όμως δεν είναι δυνατόν διότι δεν υπάρχει η τυποποίηση, δεν είναι αρκετά μεγάλες ή αρκετά μικρές οι περιφερειακές ε, ε, οργανώσει, εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση. Έχετε υπόψη τέτοιου είδου ε, προβλήματα και έχετε πάνω απ' όλα κάποια λύση σε αυτά. Απάντηση ο κύριο Κλειπ. Ναι, Όντω, <laughs> το ΑΕΠ έχει ένα πρόβλημα. Θα το πω έτσι οικό, Δεν ξέρω αν σε όλη την Ευρώπη συρρυκνούται. Εν πάση περιπτώσει όμω αυτό θα έχει όντω ε, αντικτύπωση στον προπολογισμό. Θα μα πούν δηλαδή κάποια στιγμή τα κρατη ότι είναι λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για το δε λεγόμενο non-paper από τους λεγόμενους ε, εμπειρογνώμονες που δούλεψαν υποτίθεται για τον Παρόσο. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον σε κυβερνητικό επίπεδο, ανώτατο επίπεδο αξιωματούχων δηλαδή δημόσιων υπαλλήλων, ίσως αν θέλετε διμερός και κατηδία να σας εξηγήσω περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ε, άτομα τα οποία πιέζουν για επανεθνικοποίηση, είναι που θέλουν, αυτοί που θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον προπολογισμό της Ένωσης εδώ και χρόνια και το βλέπω και στη δική μου την πατρίδα. Και τη, τελευταία ευκαιρία που το με τη Βρετανική Προεδρία όταν ε, ελήφθη η απόφαση τελικά η Μέρκελ ήταν εκείνη η οποία πάτησε πόδι. Ξέρετε τι είδους συστήσεις διαμέρισαν. Επίσης, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα βρίσκονται στο παρασκήνιο και ακόμη προσπαθούν να πιέσουν για επαναθνικοποίηση και για περιορισμό του κοινοτικού προπολογισμού, για διάθεση λιγότερων κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρόβλημα για την περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι, μια ομάδα ατόμων, ιδιαίτερα από τι ομάδε ε, ε, που έχουν μόνο εισφορά στον κοινοτικό προπολογισμό, από τι χώρε που έχουν μόνο εισφορά στον κοινοτικό προπολογισμό. Για δε την ενεργειακή πολιτική, για να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν αποκεντρωθεί η ενεργειακή πολιτική και προσεγγίσει ο καθένα με διαφορετικό τρόπο την ενεργειακή πολιτική, θα έχουμε διαφορετικέ εξελίξει προ την περιφερειακή πολιτική, την ανάπτυξη τη από την απασχόληση. Και άρα θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Γιατί, Γιατί ε, αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση με την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη τη δημιουργούμε, την εξασφαλίζουμε χάρη στις εργασίες. Στις εργασίες τις χρησιμοποιούμε χάρη στην τοπική διακυβέρνηση, στο, στη, μικρομεσαία επιχείρηση. Εκεί όπου μπορεί να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία. Κάποιο ξύπνιος που θα κάτσει κάτω και θα πει ας φτιάξω μια εταιρεία για να παράγω αυτό και εκείνο. Όχι από κάποιο κράτος που θα τους δώσει μια εντολή σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί από τη μια μικρομεσαία επιχείρηση προκύπτει μια άλλη, βρίσκεται δουλειά για μια τρίτη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα τομέα τη ενέργεια, σε παραδείγματι, που μπορούμε πραγματικά πολλά να κερδίσουμε και να προσφέρουμε. Περιβάλλον και ενέργεια. Μένα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζουν από την περιφερειακή πολιτική ή από ποια άλλη πολιτική. Και αν θέλουμε να κρίνουμε, πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώ τι έχει δαπανηθεί σε κάθε περίπτωση. Ανατολική Ευρώπη, ναι. Δεν ξέρω αν, αποτελεσματικό το, αν είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε. Τώρα λίγο κατάλαβα τι εννοούσατε. Ε, το κρίσιμο σημείο, πιστεύω, είναι ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής των τοπικών αρχών, αρχόντων από την Πολωνία Φερρυπίν ακούω ότι θέλει η πολωνική κυβέρνηση να αναθέσει περισσότερε εξουσίε, να εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες περιφέρειες, να διαθέτει περισσότερα κονδύλια ε, για διαχείριση στις ε, περιφέρειε, Αλλά για να σα δώσω ένα παράδειγμα από άλλη χώρα, τη Σερβία, την οποία πρόσφατα επισκέφθη, που έχει πολύ κεντρική οργάνωση, μία ε, περιφέρεια ουσιαστικά με την Βοηγοδίνα στο βορρά, όλα τα υπόλοιπα εργαζόμενται κεντρικά από το Βελιγράδι. Μα κάλεσαν λοιπόν δήμαρχοι από την Ανατολική Σερβία, οι οποίοι μας είπαν, εμείς οι δήμαρχοι, κάτσαμε κάτω, από διάφορα κόμματα, κάτσαμε κάτω λοιπόν μας λένε και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε μια ε, υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί η απόφαση και βέβαια σε ένα βαθμό και από το Βελιγράδι, αλλά πάνω απ' όλα από εμά. Ε, γιατί αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάρουμε τη μοίρα μα στα χέρια μα, γιατί το Βελιγράδι ποτέ δεν θα μα βοηθήσει να εξασφαλίσουμε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Ε, μόνο εμεί οι περιφερειακέ αρχέ μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και όταν του ρώτησα αν έχουν κάποιο κοινό θέμα, κάποιο κοινό πεδίο, η απάντηση ήταν. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό, γελάσαν όλοι. Είμαστε όλοι πανάπτυκτοι. Όλη η Ανατολική Σερβία. Αλλά βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν πουλάει πολύ στην κεντρική εξουσία. Γι' αυτό ανέλαβαν μόνοι του την, ε, την, πρωτοβουλία. Τέτοιου είδου πολιτικέ, τέτοιου είδου περιπτώσει ασφαλώ μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα. Ε, Επίση, ε, προσβασιμότητα στα κονδύλια. Σύντομη απάντηση, υπάρχει μια ομάδα ανώτατου επίπεδου για το γραφειοκρατικό φόρτο που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο επιτροπή και ο Μπαρόσο από τον προηγούμενο μα ε, πρόεδρο, από τον Ρικάρδο Ήλι, είχε ζητήσει να λάβει μέρο σε αυτή την ομάδα του επίπεδου. και φαίνεται ότι θα πάει καλά αυτή η ομάδα. Δεύτερον, εμεί στη δική μα οργάνωση, στη Γενική Συνέλευση, λάβαμε την απόφαση για σύσταση μια ομάδα εργασία η οποία θα παρακολουθεί του διάφορου μηχανισμού χρηματοδότηση, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή ε, γίνεται η διαχείριση τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα επανέλθουμε για να σα μιλήσουμε, γιατί εσεί δυστυχώ είστε ο μόνο σύμμαχο που έχουμε. Ο μόνο σύμμαχο ο οποίο μπορεί να εξασφαλίσει, μπορεί να ελέγξει ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι γενικέ Διευθύνσει, τα διαφορετικά προγράμματα διατίθεται με τρόπο ευχερή, χωρίς δυσκολίε. Για να μιλήσω για τον πόντο, τον εύξηνο πόντο, έχουμε περιφέρειες από την Ανατολική Γειτονία, εταιρική σχέση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μελλοντική, πώ το λένε αυτό, προενταξιακή βοήθεια, διάφορου δηλαδή κλάδου. Ε, με διάφορου κανόνε, διαφορετικού κανονισμού, στου οποίου υπάρχει το κάθε κονδύλιο και είναι πολύ δύσκολο. Όποιο θέλει να πάει να αναπτύξει δραστηριότητε σε επίπεδο ε, εύξηνου πόντου, είναι αδύνατο να βρει άκρη. Γι' αυτό λοιπόν εμεί θα κάνουμε τη μελέτη μα θα... και θα επανέλθουμε ασφαλώ με νέε προτάσει σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει, κυρία Χιούπνερα, εκ μέρου των συναδέλφων όλων μπορώ να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα τη ε, Συνέλευση των Περιφερειών τη Ευρώπη για την ανταλλαγή αυτή απόψε αγαπητοί συνάδελφοι. Ασφαλώς ε, σας εκφράζω όλους λέγοντας ότι και εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας με την ε, συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και περιμένουμε να σας ξαναδούμε και να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων, ε, να ενημερωθούμε από εσά, να εμπλουτιστούμε από την εμπειρία σας και από ποια άλλη τεκμηρίωση έχετε ενδεχομένω και φυσικά να έρθουν σε επαφή συναδέλφοι μέσα ο κύριος Κλίπ. Βεβαίως παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας ε, με μένα ή με τους συναδέλφους μου. Μπορείτε να μας βρείτε ε, με τα αρχικά αε ρο, A-E-R, Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Assembly of the European Regions, και από εκεί μπορείτε και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο και απευθεία επικοινωνία, ε, διεύθυνση ταχυδρομική κτλ. να βρείτε. Η κυρία Χιμνερ, ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε που σα διακόπτω έτσι γιατί έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημείο 5. Ελπίζω να είναι εδώ κύριο Κυρίλοφ. So I would like to just remind us that we are uh, now there is. Uh, λοιπόν, ε, ξέρετε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, θα έλεγα, που έχει να κάνει με τη θέση σε ισχύ ε, τη συνθήκη Λισαβόνα από την 1η Δεκεμβρίου. Επειδή έχουμε κρεμεί ε, κανονισμό και έδωσε και ο Λαμπέρ ένα άλλο παράδειγμα, εδώ είναι πιο πολύπλοκό το ζήτημα και θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από τον κύριο Κύριλοφ και στη συνέχεια θα ήθελα να κάνει και ένα σύντομο σχολιασμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού βρισκόμαστε και πώ θα βγούμε από την κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί έχουμε καθυστερήσει. Θα ήθελα να ακούσουμε και την άποψη όμω των συναδέλφων της Επιτροπή. Γιατί όπως είπατε, η κατάσταση περιπλέκεται. Και σήμερα δυστυχώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε την ουσία, αλλά άλλα ζητήματα. Και δεν είναι η πιο τυχερή μου αποστολή θα έλεγα, αλλά τι να κάνω. Τα έγγραφα εργασία προετοιμάστηκαν για λόγους ε, διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή διαδικασίας και τις πρόσφατες εξελίξεις. Από συγκατάθεση πάμε στη συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή εφαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Ε, yes, this procedure, as you know... Μάλιστα, επαναλαμβάνω. Όπως ξέρετε, αυτή η διαδικασία αναγνωρίζει νέε αρμοδιότητε στο Κοινοβούλιο και δυνατότητα να επιδράσουμε απευθεία στο τελικό αποτέλεσμα. Όμω εδώ πρέπει να απαντηθούν ορισμένα πρακτικά νομικά ζητήματα. Πριν αρχίσουμε, πρακτική φύση, να αρχίσουμε με την ουσία. Πρώτα, από πότε επίσημα θα δίνει τη ε, γνώμη του το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα στείλει μία omnibus communication με κατάλογο όλων των εκκρεμών προτάσεων που καλύπτει η νέα αλλαγή και θα προτείνει και τη νέα διαδικασία. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσημα να εργαζόμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεύτερον, ποια πρόταση θα αποτελέσει τη βάση για την εργασία στην Επιτροπή. Πρέπει να, ξε... να σας πω ότι εδώ έχουμε πάρει αντικρουόμενα μηνύματα. Πρόσφατα κάπως και καθαρίζει το τοπίο. Είτε το αρχικό κείμενο της Επιτροπής με ημερομηνία 22 Ιουλίου ή μια νέα πρόταση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, θα ε, πρόκειται για το αρχικό κείμενο. Επίσης, η πρόταση θα αποσταλεί και στα εθνικά κοινοβούλια. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Πάντως ξέρουμε την άποψη των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, που η απάντηση είναι ναι. Τέταρτον, Όσον αφορά τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή απασχόληση, ποια θα είναι η απόφαση. Δεν ξέρω αν ξέρετε συνάδελφοι, έχει ζητήσει ε, να είναι κύρια ε, Επιτροπή επί τη ουσία η Επιτροπή απασχόληση. Ή τουλάχιστον ε, να έχει μοιραστεί από κοινού τι αρμοδιότητε μαζί μα. Και τι θα γίνει με την απόφαση αυτή λοιπόν για τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Μόλις έχουν ξεκαθαριστεί όλα αυτά τα στοιχεία, και θα έχει δώσει ε, και την γνώμη του Κοινοβούλου, τότε θα αρχίσει η εργασία επί Λυπάμαι, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα αρχίσουν σύντομα. Και δυστυχώς όλα αυτά τα μέτρα είχαν ε, ως σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι μόλις συμπεριλέψουμε όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα θα έχει τελειώσει και η κρίση. Υπό το φως της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, ε, κάτι γίνεται με το μικρόφωνο από ό,τι φαίνεται. Sorry. συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε πολύ αργότερα, μετά το Γενάρη. Τώρα θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Για να καταλάβω σε γενικές γραμμές τι πιστεύετε και να προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε τι θα γίνει συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με τη, με τη θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Είναι όμως πολύ σημαντικό οι τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού να εγκριθούν ως δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ακριβώ αυτό το νόημα έχει η απλοποίηση της νομοθεσίας. Να βοηθηθούν οι χώρες ε, εν καιρό κρίσης και όχι μετά θάνατον. Δεύτερον, είναι προφανές ότι η καθυστερημένη έγκριση των αλλαγών θα μας οδηγήσει σε μια πολύ καθυστερημένη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, τις επιπτώσεις της κρίσης, κυρίως οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Με βάση την απόφαση Κορεπέρ πρέπει να πιέσουμε τα πράγματα για να προχωρήσουμε με βάση τη συμφωνία που έχουμε. Η ε, νέα πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σημαίνει ότι πάμε προ τα πίσω αντί προ τα εμπρό. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει ε, πρέπει ε, να βρούμε μια λύση προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειαζόμαστε και θέλουμε να υλοποιηθούν αυτές οι διατάξεις το πρώτο εξάμεινο του διο... Ε, το πρώτο μέρος του χρονικού διαστήματος 2007-2013, δηλαδή τώρα. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν παράλογη και θα αποτελούσε ήττα και της δικής μας Επιτροπής. Τέλος για τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την Επιτροπή Απασχόλησης, είναι σαφές ότι ε, αυτό το θέμα είναι τελείως αβάσιμο. Και αν επιτρέπετε να είμαι κοινικός, ίσως ο μοναδικός λόγος είναι η καθυστέρηση των μέτρων αυτών, έτσι ώστε να έχει τελειώσει η κρίση. Και πλέον δεν θα είναι απαραίτητα τα μέτρα αυτά. Γι' αυτό ελπίζω η συνδιάσκεψη των Προέδρων, κυρία Πρόεδρε, ε, απευθύνω σε εσά προσωπική έκκληση. Έτσι ώστε στην διάσκεψη των Προέδρων να λάβει την σωστή απόφαση. Ήταν άδικο και δεν μπορέσουμε να το εξηγήσουμε σε κανένα Ευρωπαίο πολίτη. Δηλαδή αποτύχαμε μόνο και μόνο λόγω κάποιων γραφειοκρατικών και νομικίστικων εμποδίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιεροκόνη. Madame Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πω τίποτα άλλο όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Ε, είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας και όσον αφορά το κείμενο που θα μας δοθεί, αλλά και όσον αφορά την ημερομηνία στην οποία θα δοθεί. και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μποστινάρου. στόχο ήταν να βοηθηθούν οι χώρε που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και τι περισσότερε δυσκολίε ε, στην παρούσα κρίση. Και τελικά, λέει η κυρία Μπριάρο Κονή, δεν θα τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά ε, ε, και θα τελειώσει η κρίση. το ΕΛΚ εξακολουθεί να συζητά την ομόφωνη συμφωνία στο Συμβούλιο και τώρα πρέπει να δούμε βεβαίως κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία. Πάντω, το θέμα είναι ότι μόλις, αυτές, μόλις ξεπεραστούν αυτές οι βεβαιότητες πρέπει να δράσουμε ιδιαίτερα γρήγορα. Όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με την έναρξη ισχύω της συνθήκη της Λισαβόνας και με, ε, ε, και με την θετική πορεία για τη δημοκρατία. Όλοι θα πρέπει όμως να δράσουμε γρήγορα ε, για την οικονομική κρίση που επιδρά αρνητικά στους πολίτες και στι επιχειρήσει. Θα έχουμε δύο μήνε προβληματισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου χρονικού διαστήματο θα ζητήσουμε την άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Α ε, αξιοποιήσουμε αυτού του δύο μήνε για να εργαστούμε. Αλλά να προσέξουμε το εξή. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν θα πρέπει να επιβραδύνει τι διαδικασίε για τόσο σημαντικά ζητήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με την ε, υφιστάμενη κρίση. Ήδη ε, είπα στον εισηγητή ότι ε, είμαι στη διάθεσή του. Σας επιβεβαιώνω ότι είμαι έτοιμη ε, να συναντηθώ με τους άλλους όλους εισηγητές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα που αποτελούσε και αρχική πρόθεση. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο γρήγορα και η εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας, όπως είπα, να μην ανακόψει αυτή την απόφασή μας. Ο κύριος Λούχαν. Vă Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω και εγώ αυτά τα οποία είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Πρέπει να αρχίσουμε την τροπολογία του κειμένου της Επιτροπής τώρα. διαφορετικά δεν πρόκειται να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έξοδο από την κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί... Ε, έχουμε παρόμοιες απόψεις παρά τις ε, αντίθετες πολιτικές ομάδες στις οποίες ανήκουμε. Υποστηρίζω λοιπόν και την άψη του κυρίου Μποστινάρου. Το θέμα είναι ε, ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να πλησιάσουν πιο κοντά ε, τους ευρωπαίους πολίτες. Και αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική, κυρίως για τα καινούργια κράτη-μέλη. Θέλουμε την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, μα ήδη έχουμε καθυστερήσει πρέπει να ξεκινήσει όλη η διαδικασία αμέσως σε επίπεδο δικής μας Επιτροπής και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες όλων των μελών της ομάδας. Ευχαριστούμε, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Γκοντμάνης. Εγώ θα... Ε, ε, έχω διαφορετική άποψη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πλήρες μέλος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και για δύο μέρες συζητάγαμε ε, την κατάσταση. Σήμερα είχα τη δυνατότητα να εξηγήσω την πραγματική κατάσταση ε, στο, ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ωραία, αντί να μιλάμε για τι τυπικότητε, θέλετε να μιλήσουμε για την ουσία. Εντάξει, θα είμαι σύντομο. Δείτε το ε, κοινωνικό ταμείο από τις, κάτω από την προηγούμενη προοπτική, δηλαδή χωρίς την κρίση. Δεν θα, δεν θα κατανομάσω χώρες, γιατί, για λόγου διοντολογίας. Αλλά να σα πω ότι στο διάστημα 2000-2006 έπρεπε να έχουμε να φτάσουμε στο 95% ως ρυθμό πληρωμής. Δηλαδή ε, χρήματα που πληρώνονται αναδέσμευση. Αντί όμως για το 95, πολλές χώρες έφτασαν στο 83, 73, 81 και ο ρυθμός πληρωμών ήταν πολύ ε, ε, χαμηλότερος και πριν από την κρίση. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, έτσι. Και πολλές χώρες που ε, εκπλήρωσαν το στόχο του 95%, ναι, ήταν αρκετές. Άρα, αλλά να δούμε το εξή. Η διαφορά αυτή είναι μεγάλη. Αυτό όμως δεν οφείλεται στη γραφειοκρατία των ευρωπαϊκών θεσμών. αλλά δεν ήταν παρόμοιος ο ρυθμός συμμόρφωσης, δηλαδή υποβολή των κατάλληλων εντύπων κτλ. Τα... Γύρω στα 16 δις δεν εδόθησαν από τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Περιλαμβάνεται και το Ταμείο συνοχή τα κονδύλια για τη συνοχή. Γιατί πρέπει να δοθούν τα, έπρεπε να δοθούν τα έγγραφα μέχρι το τέλος του 2010. Αλλά αν μιλάμε όμως για το κοινωνικό ταμείο, τα, οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερε από ό,τι θα έπρεπε. Και τώρα, μιλάμε για τις νέες προοπτικές, έχουμε τα, πιο πρόσφατα αποτελέσματα, τα οποία είναι δυνατόν να τα πάρουμε. Και θα δείτε σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τι πιο πρόσφατε πληροφορίε, το κοινωνικό ταμείο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Ξεκινάμε από 13% ρυθμό πληρωμής μέχρι 50%, δηλαδή 4,5-5 φορές διαφορά. Και για λάβετε υπόψη και την κρίση και ε, εξετάστε τις διαφορές και από άψη ΑΕΠ. Θα δείτε δεν υπάρχει σχέτιση. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτοί που βρίσκονται στην κρίση δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν κάτι τέτοιο. Και τέλος. Κοιτάξτε, σήμερα ξε, τελειώσαμε 122 δις ε, για πληρωμές. Τελειώσαμε λέει, όλο τον ολοκληρωμένο προπολογισμό. 120 έδωσε το Συμβούλιο. Ε, ε, όλα τα καλύψαμε μέσα. Κοσλοντούι και τα λοιπά. Αλλά δεν υπάρχουν άλλα χρήματα από το 2010. Σήμερα τελειώσαμε. Αν, αν μιλάμε για 6,6 σε 2 χρόνια, 3 το 2009, 3 το 2010, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Το περιθώριο είναι σχεδόν μηδέν. Ε, άρα μπορούμε να ξαναπάμε στα κράτη-μέλη και να ρωτήσουμε. 6,6 ακόμα θέλετε που ζητήθηκε να δοθούν ε, με 100% ε, επιστροφή από τα κράτη-μέλη. Μα δεν είναι εύκολο. Σύμφωνα με τον προπολογισμό του 2009, ακόμα 20 μέρες έχουμε αυτό το τέλος. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστικοί. Δεν θα λυθούν τόσο εύκολα τα προβλήματα. Και δεν έχει νόημα και εμεί να πιέζουμε. Το ζήτημα είναι το εξή. Α, και κάτι τέλ. Άρα, τελευταίο. Τότε μιλάμε για δάνειο. Άρα θέλουμε ένα, ένα όργανο, ένα θεσμό που να παρακολουθεί το δάνειο. Και το 2011, 2012, 2013 οι πληρωμές θα μειωθούν, γιατί έχουμε υπερπληρωμές το 2009-2010. Οπότε έχουμε πάρα πολλά προβλήματα γιατί έχουμε τα επιτόκια, ε, πρέπει να αντληθούν τα κονδύλια και το βασικό θέμα είναι το εξή. Ή τώρα είναι πολύ αργά γιατί δεν είμαστε μέσα στον προπολογισμό και δεύτερο, σα ζητώ συγγνώμη, αλλά αν δούμε τα θέματα αναχώρα θα δείτε πολύ εύκολα ότι ε, η υλοποίηση, η συμμόρφωση και πριν από την κρίση ήταν τόσο διαφορετική, σας το είπα, δεν έχει καμία σχέση με την κρίση. Ε, έτσι κι αλλιώ ε, υπήρχε πρόβλημα με το κοινωνικό ταμείο, ακόμα και με το ταμείο συνοχή. Η, η, η διαφορά είναι 4-4,5 φορέ ε, σε σχέση με σήμερα. Υπάρχουν χώρε που βρίσκονται κάτω από το 10%. Ορισμένε είναι στο 16% και άλλε στο 60%. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται και να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτά τα προβλήματα, να αναλύσουμε προσεκτικά τα αριθμητικά στοιχεία ή να φτιάξουμε μια ομάδα εργασία με την δική μα Επιτροπή και με την Επιτροπή Προπολογισμού, γιατί αυτό το θέμα αφορά και τι δύο επιτροπέ. Πάντω δεν είναι εύκολο. Και η Επιτροπή Προπολογισμού θα μα ρωτήσει, θα ρωτήσει, θα ζητήσει την Επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσει. Τι θα συμβεί με τα κονδύλια τα οποία δεν καταβλήθηκαν γιατί οι χώρε δεν εκπλήρωσαν τα κριτήρια. Ή θα μεταφερθούν ή δεν θα πληρωθούν καθόλου. Συμπεριλαμβάνοντα και τι πληρωμέ για το κοινωνικό ταμείο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν μπορούμε διαρκώ να πιέζουμε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να κάνει το Α ή το Β. Γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Σα ζητώ συγγνώμη για αυτέ τι πληροφορίε που σα δίνω τώρα. Ε, όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τη δική μου η οποία αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τη διαδικασία διότι δεν είναι σαφές ε, πάντα το τι έπρεπε να έχει γίνει και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τι συνέβαινε, ότι με βάση την παλαιά διαδικασία, διαδικασία της ε, ε, σύμφωνης γνώμης, σήμαινε ότι το Κοινοβούλιο έκανε μία γνωμοδότηση με εντολή για τον ε, διαπραγματευτή του άτυπα να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει όμω ούτε από του διάσκεψη των Πρόεδρων, ούτε από τον εισηγητή. ω του εντολή για τον εισηγητή δεν υπάρχει. Μέχρι σήμερα. Άρα, στη διαδικασία αυτή το κοινοβούλιο δεν έχει αξιοποιήσει τις πραγματικέ εξουσίε που έχει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Οπότε το, ο κίνδυνο είναι ότι είτε θα λάβει εντολή ο εισηγητή, που μέχρι τώρα δεν έχει εντολή για την πραγμάτευση, μόνο συζητήσει έχει παρακολουθήσει διότι δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν, γιατί ακόμη και με την παλαιά διαδικασία δεν υπήρχε αυτό το δικαίωμα. Τώρα στην πράξη, όντω υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, υπάρχει κορεπέρ, υπάρχει απόφαση του κορεπέρ και το ερώτημα που είναι πώ προχωρούμε από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε τουλάχιστον ότι έστω δεν υπάρχει πρωτοβουλία της Επιτροπής, αλλά το Συμβούλιο έχει μόλις ολοκληρώσει μια ανάγνωση και έχει καταλήξει σε μια θέση. Όμως το Κοινοβούλιο δεν έχει θέση. Η Επιτροπή μας δεν έχει θέση. Δεν υπάρχει εντολή για τον εισηγητή μέχρι σήμερα. Και το ελάχιστο που πρέπει να επιτύχουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί, να προχωρήσει μια διαδικασία μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα στην Επιτροπή μας, με την οποία θα διατεθεί εντολή, θα προκύψει εντολή για τον εισηγητή, αλλιώς θα έχουμε ουσιαστικά απεμπολίσει τις εξουσίες μας και γι' αυτό πρότασή μου είναι, ανεξαρτήτως της διελκυστίνδας εδώ, για το κατά πόσο να ακολουθούμε την παλαιά ή τη νέα διαδικασία. Εγώ προτείνω συγκεκριμένα να επιδιώξουμε μια διαδικασία, να ξεκινήσουμε στην Επιτροπή μα μια προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, με μια έκθεση από τον εισηγητή και όχι μόνο ένα έγγραφο εργασία, αλλά έκθεση του εισηγητή, βάσει του οποία θα μπορούμε μετά να πούμε, να συζητήσουμε εάν μένουμε στην έκθεση πρωτοβουλία ή εάν ε, προχωρούμε σε κλασική μορφή έκθεση. Αυτό. πρόθεσμα μέσα στις 8 εβδομάδες που έχουμε, ένα, μια, ένα περιθώριο και για τα εθνικά κοινοβούλια και επιπλέον τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρόνο γιατί μπορούμε να δουλεύουμε παράλληλα. Νομίζω ότι αυτές τις 8 εβδομάδες μπορούμε ως προθεσμία να τις στηρίσουμε. Είναι ρεαλιστικό. Με βάση το έγγραφο του Κορεπέρ. Ή Μπορούμε να πούμε στο ε, Συμβούλιο ότι τελικά αυτό το παλιό έγγραφο της Επιτροπής έχει τροποποιηθεί από το Κορεπέρ, ότι γνωρίζουμε πως η Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα έχει την ε, πρόθεση να ακολουθήσει για τη νέα της πρόταση το έγγραφο της Κορεπέρ, θεωρείται δεδομένο αυτό. Και άρα ας πάρουμε και εμείς ως βάση το Κορεπέρ, το έγγραφο του Κορεπέρ που θα αποτελέσει θεωρητικά και τη βάση για την πρόσθεση επιτροπή. Με βάση αυτό το έγγραφο του Κορεπέρ παίρνουμε μια απόφαση και την εντολή για τον εισηγητή. Αυτό είναι το καθήκον μα. Αυτό είναι το καθήκον που δεν έχουμε ακόμη επιτελέσει. Εντολή λοιπόν πρώτα απ' όλα. Και μετά να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, εάν θα πρέπει να περιμένουμε να εκπνεύσουν οι 8 εβδομάδε πράγμα που θα προτιμούσα εγώ για να είμαστε και σίγουροι ότι όλα έχουν τηρηθεί όπως πρέπει, αν και δεν έχουμε αρκετό χρόνο, μέχρι την αποφασή σε επίπεδο και από την Επιτροπή και μέχρι την Ολομέλεια μπορούμε να το ξανασκεφτούμε και να δούμε αν θέλουμε να έχουμε μια πιο τυπική μορφής απόφαση ως προς την τήρηση των διατάξεων συνθήκης Λισαβόνας, αν εφαρμόζονται δηλαδή αυτές ή όχι αλλά ακόμα δεν είναι σε φύση κατάσταση. Δεν υπάρχει απόφαση τη επιτροπή μα, δεν υπάρχει συζήτηση μέσα στην Επιτροπή μα μόνο διαδικαστικά ζητήματα έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμή. Επί του ουσία τίποτα. Ανεξαρτήτως όμω τη διαδικασία που θα επιλέξουμε, πρέπει εμεί τώρα να διαλέξουμε, να ξεκαθαρίσουμε ποια προθεσμία θέλουμε για τι τροπολογίε, πώ θα λάβουμε την απόφαση μέσα στην Επιτροπή μα, να προχωρήσουμε στην απόφαση αυτή για να δώσουμε εντολή στον εισηγητή. Γιατί μέχρι τώρα ο ονόματο μόνο διαπραγματεύεται και όχι εξ τη Επιτροπή μα. Επαναλαμβάνω, ούτε μία φορά δεν έχουμε μπορέσει να ε, συζητήσουμε την εντολή και να λάβει υπόψη του εισηγητής επίσημος εισηγητής επισήμως των σκιωδών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με την προλαλή σα, όπως επίσης και, ε, και με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ε, ω προ τα δικαστικά και, και τη σημασία του θέματος και λόγω της σημασίας του θέματος νομίζω ότι θα πρέπει να χώσουμε το ποδαράκι μας στην πόρτα και ε, να μπούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία. Έχουμε στόχους που πρέπει να είναι ξεκάθαροι το ταχύτερο δυνατό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό λόγο υπάρχει για μένα. Να μπορέσουμε να έχουμε το ταχύτερο δυνατό στοιχείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι ώστε εάν κάτι δεν πάει καλά να είμαστε θέση να παρεμβαίνουμε αμέσως. Και για, το, και να μπορούμε να παρακολουθούμε το γραφειοκρατικό φόρτο και τις λοιπές συνθήκες που επικρατούν. Σε αυτό το σημείο ακριβώ νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε με προσοχή πώς παρακολουθούμε ε, σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις. Και βέβαια ανάλογα με τις συνθήκες της Λισαβόνας, ε, εάν θα φορμούν διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας ή όχι. Νομίζω κανείς άλλος συνάδελφος δεν θέλει τώρα το λόγο ή κάνω λάθος. Α, με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Οκονή. Όσον αφορά την Κομισιόν και τον φάκελο FSE, εκτός αν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι ένα μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας που ζήτησε η Κομισιό να ασχοληθεί με αυτό το φάκελο. Ίσως λοιπόν μπορείτε να συζητήσετε μέσα στην ομάδα σας για να επισπεύσουμε. Ίσως μπορείτε να αποσύρετε δηλαδή το αίτημα που υποβλήθηκε για να εξεταστεί ειδικότερα από την Κομισιόν το, το τμήμα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, λέει η Πρόεδρος, ότι έχω απαντήσει στην επιστολή της κυρίας Περβάνς Και η συνδιάσκεψη των Προέδρων δεν μπορεί να λύσει αυτό το θέμα προτού ξεκινήσει η διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το κανονισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή τη φάση. Λυπάμαι. Λοιπόν, Τώρα θα ήθελα να ζητήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να μας ενημερώσει για το πού βρισκόμαστε από την άποψη της Κομισιόν αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν ετοιμάζει την απόφαση για το Omnibus, όπως λέγεται. Θα είναι στο τέλος της ημέρας έτοιμη και θα έχουμε εξηγήσει και για αυτό το φάκελο τι γίνεται με βάση αυτή την απόφαση Omnibus. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω τη γραμμή των νομικών μας υπηρεσιών. Είναι η εξή. Κατά την άποψή τους, η Κομισιό έχει ήδη επισήμως διαβιβάσει στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούλιο βάσει της διαδικασίας τυπικής έγκρισης την αρχική πρόταση Συνεπώς δεν χρειάζεται να υποβληθεί άλλη πρόταση από την Κομισιόν. Δεν απαιτείται αυτό. Καθώς δεν υπάρχει και τυπικά νέα πρόταση που να έχει προκύψει. Όμως, οι νομικοί μας επίσης τονίζουν ότι ε, από τότε δημιουργήθηκε μια πολιτική πραγματικότητα στο Συμβούλιο, η οποία οδήγησε σε ένα ενδιάμεσο βήμα μέσω ενός non-paper της Κομισιόν, με το οποίο υποβλήθηκε μία πρόταση ε, παρόμοια με αυτήν που εγκρίθηκε ομόφωνα στο Κορεπέρ. Συνεπώς τώρα, επειδή το πολιτικό, έχουμε σαν πολιτικό γεγονός την απόφαση του Κορεπέρ. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτήν θα συνεχίσουμε την εργασία μας. Ωραία. Φαίνεται όμως να υπάρχει ένα νομικό ερώτημα, ε, ερωτηματικό μάλλον, για το κατά πόσο το Συμβούλιο μπορεί επισήμως να διαβιβάσει αυτή την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θα ληστεί στο επίπεδο του νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, δηλαδή κατά πόσο μπορεί για τυπικούς λόγους να διαβιβαστεί αυτό το έγγραφο στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε κατά τα λοιπά, η Κομισιόν δέχεται αυτή την απόφαση του Κορεπέρ σαν πραγματικότητα. Και είναι προς συμφέρον των θεσμικών οργάνων να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν ώστε να απλουστεύσουμε τα μέτρα και να προχωρήσουμε στα δημοσιονομικά μέσα που προβλέπονται για τις διάφορες χώρες το ταχύτερο. Κατά την άποψή μας, δηλαδή, αυτό το οποίο θα εμφανιστεί, τα προκύψει μάλλον, και εδώ έχουμε τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου σαν κινητήρια δύναμη μέσα στη διαδικασία της συναπόφασης, Έλεγα λοιπόν ότι εμείς αναμένουμε ε, το υπόλοιπο της εργασίας να πραγματοποιηθεί με ένα τρίλογο, ο οποίος θα ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν. Πρόεδρος. Έχετε ερωτήσεις προς την Κομισιόν, θέλετε άλλες διευκρινήσεις ίσως ή είμαστε εντάξει. Εξ όσων λοιπόν καταλαβαίνω, η κατάσταση έχει ως εξής. Πρέπει να λάβουμε το παραπεμπτικό για να ξεκινήσουμε τυπικά. Αλλά έχουμε συμφωνήσει πριν ένα μήνα και πριν από δύο μήνες έχουμε συζητήσει τις διαδικασίες και έχουμε ε, συμφωνήσει να άτυπα να προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με την άτυπη εργασία ώστε να μην καθυστερούμε όλοι, όλες τις διεργασίες περιμένοντας την έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβουλία. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι συνάδελφοι που πήραν το λόγο τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της εργασίας βάση ε, τη, του Κορεπέρ, χωρίς να ξέρουμε τι η Κομισιό ή το Συμβούλιο θα στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλό είναι αυτό, διότι οι εισηγητές έτσι μπορούν να ξέρουν προς τα πού να κατευθυνθούν συντάσσοντας την έκθεση. Αλλά τυπικά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας πριν λάβουμε το παραπεμπτικό από την Ολομέλεια. Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται πώς θα περάσει και τυπικά η πρόταση προς το Κοινοβούλιο. Θα βρεθεί η λύση, θα εφαρμοστούν οι διάφορες διαδικασίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Α, κάποιο. Η κυρία Σάτεν ζητά το λόγο. Λίγο πολύ αυτό που είπα και πριν. Ένα πρόβλημα παραμένει ανεπίλητο ακόμη, ότι δεν έχει τοποθετηθεί για το έγγραφο αυτό η Επιτροπή μας μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει εντολή για τον ε, εισηγητή δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στον τριμερή διάλογο, δηλαδή το κοινοβούλιο απεμπολεί εδώ τα ε, δικαιώματά του, τις του. Και εσεί, ω Πρόεδρος θα πρέπει να μεριμνήσετε, να διαμορφωθεί η θέση της Επιτροπής μας, δηλαδή μία έκθεση με προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε ένα τριμερή διάλογο. Είναι η μόνη δυνατότητα να μπούμε μέσα στη διαδικασία. Αλλιώ είμαστε εκτό παιδιά. 100% εκτό παιδιά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαίωσει ότι τηρεί τι δικέ τη προθεσμίε και η μόνη η οποία δεν μπορεί να τη στηρίσει είναι η Επιτροπή των, των Περιφερειακών Υποθέσεων. Είναι άδικη η κρίση που διατυπώνεται όπως ξέρετε, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει λάβει το έγγραφο, το οποίο πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια. Και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Και προς το παρόν υπάρχει μια διαφορά απόψεων μεταξύ των νομικών υπηρεσιών της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, και αυτό έκανε και ο κύριος Κύριλοφ τους τελευταίους δύο μήνες, είναι άτυπα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι εμπεριέχεται στον κανονισμό, ώστε από τη στιγμή που μπορούμε επισήμω να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, να προχωρήσουμε. Και θα προχωρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να παροβιάσουμε τους κανόνες. Αλλά θα κάνουμε όλες τις απαραίτητε προσπάθειε για να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Ο, κύριο Συμφωνώ μαζί σα, κύριε Πρόεδρε. Χάσαμε το μικρόφωνο. Πανέρχεται. Βεβαίως αυτή η παραπομπή είναι απαραίτητη ώστε η Επιτροπή ε, να δώσει τις οδηγίες. Αλλιώς θα γελιοποιηθούμε θα γίνουν αστεία τα πράγματα. Δηλαδή, επισήμω δεν ξέρουμε ακόμη τι θα παραλάβουμε. Μου περάσανε κάποια μηνύματα από την Κοπισιόν την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα είναι διαφορετικά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα... Ε, δεν μπορώ να συστήσω στην Επιτροπή μα να εργαστεί πάνω σε, ένα... σε λεπτομέρειε οι οποίε είναι άγνωστε. Όταν γίνει η παραπομπή, εντάξει. Αυτή η παραπομπή δε θα χρειαστεί και υπεραιτέρω απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων αν θα οδηγηθεί στην δικιά μας Επιτροπή. Και ελπίζω ότι θα καταλήξει σε εμά και προσπαθούν και άλλοι <laughs> συνάδελφοι να βοηθήσουν γιατί πώς αλλιώς θα αναμειχθούμε. Συμφωνώ με την κυρία Σόεδρο ότι μεταξύ ανεπίσημα πρέπει να εργαστούμε, αλλά δεν φταίει η Επιτροπή. Είναι ε, το φταίξιμο είναι με το Συμβούλιο που σέρνει τα πόδια του μήνες τώρα. Και εμείς όλους αυτούς τους μήνες ε, συζητούσαμε άτυπα, αλλά δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ούτε με τα πιο απλά βήματα, εφόσον δεν έχουμε έγγραφο. Λοιπόν, καταλαβαίνω τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων, ότι όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από τη στιγμή που θα κινήσει και επισήμως η διαδικασία. Από τη στιγμή που θα φτάσει με το πακέτο Omnibus η πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο θα ενεργοποιηθούμε αμέσως και θα καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Πρόεδρος. Θεωρούμε λογικά ότι σήμερα θα αποφασίσει για το Omnibus η Κομισιό και θα έρθει άμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Δεκέμβριο η Ολομέλεια θα το παραπέμψει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος μας θα είναι να έχετε το σχέδιο της έκθεσής σας για πρώτη ανάγνωση στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, 20 κάτι νομίζω, 25 Ιανουαρίου συνεδριάζουμε μας. Να έχουμε τότε την πρώτη ανάγνωση. Ναι, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες μετά τις 8 εβδομάδες, μην ξεχάτε το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι η τελική ψηφοφορία. Εντάξει, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όλες τις προτάσεις σας τον Ιανουάριο. Κάποιος μιλάει εκτός του μικροφώνου δίπλα από την πρόεδρο. Τώρα έκλεισαν τα μικρόφωνα. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει ως προς τη μεθόδευση σήμερα λίγο πολύ. Η κυρία Σρέντερ. Πρόεδρε, εάν όντως μέχρι σήμερα. Δεν μας έχει διαβιβαστεί τίποτε. Γιατί μας λέει η Επιτροπή ότι μας έχει διαβιβάσει προτάσεις. Ας μας εξηγήσει η Επιτροπή. Εγώ δεν θέλω να κατηγορώ κανέναν άδικα. Αλλά ξέρω ότι έχουμε υπόψη μας ένα έγγραφο εδώ και καιρό και δεν έχουμε αντιδράσει. Δεν έχει ξεκινήσει το πλαίσιο της Επιτροπής μας σαφής διαδικασία. Και για το assessment, την αξιολόγηση, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε διαδικασία. Αλλά δεν το πράξαμε. θα είχε γίνει πολύ πιο εύκολη δουλειά μας, θα είχαμε δώσει εντολή στον εισηγητή, θα είχαμε μπει διαφορετικά μέσα στη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να πείτε έστω επισήμω, ναι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά εσωτερικά να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Άτυπα. Ποια θα είναι η διαδικασία, τι εντολή θα δώσουμε στον ε, εισηγητή, να του δώσουμε την ε, εντολή, να, να ορίσουμε ένα περιθώριο για τροπολογίες κτλ. Να μπορεί να κυκλοφορεί, να κάνει τις διαπραγματεύσεις του. τι φαίνεται ότι το Δεκέμβριο θα πάρουμε την ε, ανάθεση, αλλά θα πρέπει να είναι σαφής ε, η κατάσταση ως προς η εικόνα, ως προς τις τροπολογίες, ως προς την ημερομηνία δεξαγωγής της Όλα αυτά πράγματα. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω, να σας καταστήσω σας υπεύθυνη για κάποιο ε, πρόβλημα στη διαδικασία ασφαλώς όχι, αλλά παρακαλώ, επειδή η κατάσταση είναι αυτή, παρακαλώ, αναλάβετε δράση. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι, νομίζω, απαραίτητο και σημαντικό να ορίσουμε τη θέση μας, την τυπική μας τοποθέτηση για να μην χάσουμε χρόνο. Να μείνουμε εντός παιδιάς. Και να ενημερωθούμε πότε διαβιβάστηκε, όταν διαβιβαστεί, εν το έγγραφο. Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα όλες οι ομάδες. Για το αν θα παραμείνει ή όχι συγχρηματοδότηση ήταν ένα από τα μήλα της έρηδος. Ίσως θέλαμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί ως προς το να συμμετάσχουμε στη διαδικασία και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο εναργήσαμε ε, κάπως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφερόμαστε όλοι. Έχουμε όλοι διεξαγάγει τις τυπικές μας, ε, επαφ, ε, άτυπες μας επαφές. Όλοι ενδιαφερόμαστε. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε μια ευκαιρία τον Δεκέμβριο να δούμε την επίσημη θέση. Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι, εξοπλισμένοι αν θέλετε. να έχουμε μια λύση πρακτική με τον τρόπο αυτό, να επιλύσουμε τα προβλήματα και να μην ε, περιοριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις και φαινόμενα. Να κάνουμε, κατά τα φαινόμενα δηλαδή τοποθετήσεις, να κάνουμε ουσιαστική τοποθέτηση, να ξέρουμε που παρεμβαίνουμε. Επαναλαμβάνω, εγώ θα ήθελα κάποιο παράρτημα, κάποια παρατήρηση, κάποιο κείμενο από την γραμματεία, μια ενημέρωση για να παραμείνουμε ε, ενεργοί μέσα στη διαδικασία. Να μην κάνουμε το λάθος να αυτοαποκλειστούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου και πρόβλημα σε αυτό δεν υπάρχει. Μια παρατήρηση για την ε, διαδικασία και το περιεχόμενο. Όσον αφορά τη διαδικασία, 100% υποστηρίζω την πρόταση του συναδέλφου να επιταχυνθεί η διαδικασία και επίσης να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο, ε, η απόφαση του Κορεπέρ και το περιεχόμενο ναι, στη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά αν είναι πιο ευέλικτη, ευέλικτη η διαδικασία, και η συνενετική, ε, η συνεργασία, η συνενετική λήψη αποφάσεων, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις στους καλές και να αποφύγουμε τις πιο δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. Καλώ, λέει πρόεδρο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή του ταχύτερο δυνατό την διαβίβαση των προτάσεων. Παραμένει η προθεσμία για τον Ιανουάριο για να προετοιμαστείτε εσεί, κύριε Κυρίλοφ, για την πρώτη ανάγνωση. Αλλά δεν μπορούμε από τη μια μέρα να... μέχρι την άλλη να αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε τώρα δηλαδή να κρίνουμε για τη Δευτέρα. Δεν έχουμε νομική βάση. Εάν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και να προχωρήσουμε στο σημείο 6, έκθεση. Α, η Επιτροπή, το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, η Επιτροπή θα σας διαβιβάσει μόνο τη σύσταση Omnibus, η οποία εξηγεί τη διαδικασία όπως προκύπτει με την αλλαγή στη συναπόφαση. Αυτό είναι μόνο. Νέα στοιχεία, νέα έγγραφα από την Επιτροπή δεν θα λάβετε. Διότι η Επιτροπή θεωρεί ότι στις 24 Ιουλίου εφέτος διαβιβάστηκαν οι επίσημες προτάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλειωσε η υπόθεση. Το ομνεμπος απλώς επιβεβαιώνει, επαναλαμβάνει το γεγονός αυτό. Τα υπόλοιπα απλώ είναι ένα τρόπο να αντιμετωπίσουμε την πολιτική πραγματικότητα και το συμβασμό στο Κορεπέρ, όπου θεωρούμε ότι η δουλειά ουσιαστικά θα πρέπει να συνεχίσει μέσα σε μια διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Πρόεδρος υποθέτω ότι σε αυτό είναι σύμφωνη και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να μην έχουμε νέα προβλήματα. Εμείς από την Επιτροπή μας μόνο πολιτική υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε. Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά των άλλων. Can move to point number six on our agenda. Πάμε λοιπόν στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, έκτη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο τη Επιτροπή. Λοιπόν, να ζήσουμε τον Σαλβατόρε Καρόνα αν έχει να κάνει κάποια σχόλια. John, is he here? Should be. Is Mr. Carona? Yes. Mr. Carona is here. Can you just make? Grazie, Presidente. Ε, πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, για να κερδίσουμε και χρόνο. Ήδη ε, έχετε πάρει τη γνωμοδότηση, το σχόλιο δηλαδή, ε, για τη λευκή βίβλο τη Επιτροπή Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματο. Άλλωστε, την προσεχή εβδομάδα στην Κοπενχάγη, η διεθνή κοινότητα θα ε, αντιμετωπίσει το πρόβλημα ε, τη πρόθεση μια κοινή και αποτελεσματική δράση για να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει που οφείλονται στι κλιματικέ αλλαγέ. Όλοι ευχόμαστε από τη συνεδρίαση αυτή να προκύψει μια σαφής ε, και αποφασιστική, ε, για να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού ένα πρόβλημα το οποίο πλέον έχει αναγνωριστεί παγκόσμια ω η βασική πρόκληση για τις προσεχείς δεκαετίες. Πράγματι γνωρίζουμε από τώρα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της ε, ε, αλλαγής του κλίματος για τουλάχιστον 50 χρόνια. Ε, επιπτώσεις ε, που συνεπάγονται αύξηση της θερμοκρασίας της γης, ε, των θαλασσών, κίνδυνος, κινδύνους διάβρωσης των ακτών, δυσκολία εφοδιασμού τροφίμων, συνέπειες στη δημόσια υγεία, βλάβες στη βιομηχανία, στο σύστημα μεταφορών κτλ. Όλα αυτά επιβάλλουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι να λάβουμε, αποφασίσουμε μέτρα τα οποία θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων, που οφείλονται στην ανθρώπινη δράση. Δεύτερον, να προωθήσουμε μια δράση προσαρμογή που να μα βοηθήσει να ε, ε, αυξήσουμε την ε, ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής ε, πολύ σωστά ε, προσπαθεί να ορίσει ένα πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και να ενσωματωθούν οι δράσεις των κρατών μελών, να υποστηριχθούν οι πιο ε, κατάλληλες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα λοιπόν ε, να, ε, πρέπει να καθορίσουμε μια συνολική στρατηγική που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και τα μελλοντικά πιθανά σενάρια. Γνωρίζουμε ανάμεσα στα άλλα ότι η ενίσχυση ε, μια στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αποτελεί και μια τρομερή ευκαιρία, αν θέλετε, για νέες επενδύσεις πράγματι μια οικονομία ε, χαμηλής εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος που θα μας οδηγήσει σε ισχυρή ενεργειακή ασφάλεια ε, θα δώσει τη δυνατότητα να, ε, να καθορίσουμε και μια νέα ε, οδό ανάπτυξης και μάλιστα ιδιαίτερα στα σημερινά πλαίσια που διανύουμε μια τόσο σημαντική οικονομική κρίση όπως γνωρίζουμε, οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με την περιοχή και την περιφέρεια και, ε, και ανάλογα και με τα κοινωνικά στρώματα. Στην Ευρώπη ε, η Μεσόγειος ε, εκτίθεται ιδιαίτερα. Η η λεκάνη της Μεσογείου και οι όμως περιοχές και οι ορεινές περιοχές, οι ορεινές ιδιαίτερα οι Άλπεις ε, και τα νησιά, οι παράκτιες περιοχές, χωρίς βεβαίως να ε, ξεχνάμε τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες ε, περιφέρειες. Τα προσεχή χρόνια λοιπόν θα δούμε μια περαιτέρω διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης υπό αυτή την οπτική γωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον τομέα της ενέργειας οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις και στην προσφορά και στη ζήτηση. Μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε ένα σενάριο όπου ε, το λιώσιμο των πάγων, των παγετώνων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση κατά 5% της, υδροελεκτικής ενέργειας, ενώ θα υπάρξει μία μείωση τουλάχιστον κατά 25% ε, στις ζώνες της Μεσογείου. Το ίδιο ισχύει και πολλούς άλλους τομείς, ε, ε, γεωργίας, τουρισμού κτλ. Ε, δεν, θα, ήθελα, θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο ζήτημα. Αλλά και, να σα πω το εξή. Κυρίω σε μια επιτροπή όπω αυτή που έχει ω στόχο τη συνοχή ανάμεσα στι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ε, το προσέξουμε το θέμα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ε, το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις εξή πτυχές. Πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές ικανές ε, να συνδυάζουν τις δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις και να τις διοχετεύουν σε δράσεις ε, που θα μας οδηγούν σε ανάπτυξη συμβατή ε, με τις αλλαγές του κλίματος και δεύτερον και δεύτερον, να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία ε, τη Επιτροπή να, να δημιουργήσει μια συντονιστική ομάδα για τι επιπτώσει και την προσαρμογή. Ε, Τονίζοντα ιδιαίτερα ότι εδώ πρέπει να έχουμε πλήρη και ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και ευχαριστώ και του συναδέλφου για, ε, ε, για τη συμβολή του μέσω των τυχών τροπολογιών του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Στρεμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο και θα έχει, στο οποίο θα συμβάλλουμε με την ε, γνωμοδότηση την οποία συζητούμε. Η, η εισήγηση, ε, το σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορώ να πω και εγώ μερικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να παρθούν υπόψη. Ε, για παράδειγμα, ε, ε, στο σημείο 3 ε, μιλά για την ανάγκη έγκαιρης αντίδρασης στην υπερθέρμανση του πλανήτη, όχι μόνο μέσα από τα μέτρα που θα προβλέπουν περαιτέρω μείωση των εκπομπών, αλλά και μέσα από προληπτικά μέτρα κτλ. Θα ήθελα να προσθεθεί η αναφορά σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που αποτελεί και ένα βασικό αίτημα, όπως μας έχει εξηγήσει σε αντίστοιχη ερώτηση και ο Επίτροπος ο κύριος Δήμας και είναι και στην ε, κατεύθυνση δηλαδή ε, της ε, Επιτροπής. Επίσης, να προσθέσουμε στην αναφορά για τη μείωση των εκπομπών των ορίων του θερμοκηπίου το στόχο ποσοτικοποιημένο κατά 30-40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Και αυτό το αναφέρω επειδή η ε, ο μεγάλος θεσμός του IPCC μιλά για μειώσεις από 25 έως 40%. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται το 30% αν συμφωνήσουν και τα άλλα κράτη, κάτι που αναφέρεται και στην ε, Λευκή Βίβλο, ε, στην σελίδα 3. Επίσης, θα πρέπει εκεί που αναφέρουμε στα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών να προσθέσουμε το μέτρο της ενίσχυσης των δασών ε, μια και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για, και για μείωση της αποδάσωσης και για συγκεκριμένα μέτρα αναδάσωσης. Ε, θα ήθελα να προσθέσω στην παράγραφο αυτή και ε, εκεί που μιλάει για τα προληπτικά μέτρα προσαρμογής ώστε να περιοριστούν οι επιβλαβείς συνέπειές τους και μέσα μέτρα και μέσα από περιφερειακούς στόχους μείωσης της εκπομπών και περιφερειακά σχέδια προσαρμογής. Να μην μένουμε δηλαδή μόνο στο κρατικό επίπεδο. Ε, στο σημείο 5 ε, που μιλάει για τη στρατηγική ε, της προσαρμογής από το 2013 και μετά να δώσουμε έμφαση και εδώ στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές οι οποίες και απειλούνται περισσότερο από άλλες. Ε, υπάρχει επίσης, α, πιστεύω, ανάγκη στο σημείο 7 εκεί που αναφέρεται για την ε, ε, ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών με χαμηλές εκπομπών ρήπων να προσθέσουμε με έμφαση στο σιδηρόδρομο. Και αυτό ακριβώς επειδή και αποτελεί αντικείμενο, το συζητάγαμε και σήμερα το πρωί στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος, ακριβώς γιατί ο σιδηρόδρομος ξοδεύει το 1 δέκατο της ενέργειας σε σχέση με τις ε, οδικές μεταφορές. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσουμε την ανάγκη να προσανατολιστούν περισσότερο τα ταμεία συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης κλπ. προς μέτρα προσαρμογής ε, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών συμπεριλαμβανομένων αγροπεριβαλλοντικών έργων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Mr. Obermeier, please. Danke, Frau Vorsitzende. Κύριε Obermeier, πρόεδρε, ευχαριστώ η Επιτροπή αναγνώρισε σωστά ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε δύο φάσεις η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, καταρχάς, ο περιορισμός των ε, εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αφετέρου δε η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Η Αυστρία που βρίσκεται ε, κοντά στο Μόχοφσκο και το Τέμελιν, τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της Τσεχίας και της Σλοβακίας, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γεωγραφικά κιόλα και πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε μέτρα προσαρμοστικά στις ε, κλιματικές αλλαγές. Η λύση δεν Μπορεί όμω να δοθεί από του πυρηνικού αντιδραστήρε, από την πυρηνική τεχνολογία, γιατί το κόστο είναι τεράστιο, δεν έχει λυπηληθεί το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων και είναι τεράστιες πάνω απ' όλα ε, οι επιπτώσεις του οποιοδήποτε σφάλματος, του οποιοδήποτε ατυχήματος. Ένα άλλο, ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η Άλπης, ένα σημαντικό θέμα εν προκειμένου που θα πρέπει να μας απασχολήσει για να εξεύρουμε μέτρα προσαρμογής καθώς οι Άλπεις επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις κλιματικές αλλαγές με πρώιμη τήξη των πάγων, με χιονοστιβάδες ε, και ε, συρρήγνωση των παγετών νόν. Πράγμα το οποίο βεβαίως επηρεάζει και τον ε, υδάτινο ορίζοντα ολόκληρη Ευρώπης, αλλά και μεγάλους ποταμούς όπως τον Ροδανό και τον Δούναβη. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα ουσιαστικά και αποτελεσματικά γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σρότζερ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τόσο είπε ο κύριος Σόμπερ Νομίζω ότι στην γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και να δούμε ε, πώς μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής περιφερειακή πολιτική. Έχουμε παραδείγματι σημαντικό πρόβλημα με τις ε, ε, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το ζωικό κεφάλαιο. Έχουμε πολλά χρήματα τα οποία χρηματοδοτούν ε, ρηπογόνες δραστηριότητες ή επικίνδυνες για την κλιματική αλλαγή δραστηριότητες. Αναφέρθηκαν νωρίτερα και οι Άλπεις, αναφέρονται και οι παράκτιες ζώνες που κινδυνεύουν ιδιαίτερα, οι νησιωτικές περιοχές που κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε η πολιτική της συνοχής τι ρόλο διαδραματίζει, πώς επηρεάζει την κλιματική αλλαγή και πώς θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε έτσι ώστε να, αντιστρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να τις καταστήσουμε θετικές. οι τοπικές αρχές ε, από τη Ραζέτα 21 ήδη έχει αναλάβει πολύ ε, ε, σοβαρό ρόλο για την αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών, αλλά δεν έχει στην πραγματικότητα δράση ακόμη, δεν έχουν ακόμη δράσει οι τοπικές αρχές και γι' αυτό οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν στο τομέα αυτόν. Επίσης, καθήκον της Επιτροπής μας θα ήταν με τη λευκή αυτή βίβλο, με, από τη λευκή, λευκή αυτή να βρούμε σημεία στα οποία θα επισημάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδείγματα επικίνδυνα για τις κλιματικές αλλαγές ή αντίστροφα επικίνδυνα ε, παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις ως προς το κλίμα. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε μια πολύ σημαντική μελέτη Περιφέρειας 2020, όπου επισημαίνονται κίνδυνοι συγκεκριμένοι για ορισμένε περιοχές, για ορισμένε περιφέρειες. Αναφέρονται τα ποσοστά πληθυσμού που θα επηρεαστούν εάν προχωρήσει με τους ραχδαίους ρυθμούς η κλιματική αλλαγή που έχει ήδη. Τι είδου ζημία θα αντιμετωπίσουν αυτές οι περιφέρειες. Όχι μόνο η βιολογική ποικιλία, βιοπικιλία που είναι πολύ σημαντική, αλλά η ε, κίνδυνη για την επιβίωση των ίδιων των τοπικών αυτών ε, οικισμών ή ομάδων πληθυσμού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, πιστεύω, με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με της ευκαιρίας, πριν να στον Όστο Φαριστέλ Ρόι, αυτό το οποίο δεν έχει το κείμενο είναι η συνεισφορά των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι καθήκον μας να ακούσουμε προσεκτικά αυτό τα οποίο είπε η κυρία Σέντερ. Τη συμβολή δηλαδή των πολιτικών. Ρόι. Θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είμαι πλήρω ικανοποιημένο με το κείμενο. Μπορώ να σα διαβάσω διάφορα εδάφια εδώ με τα οποία διαφωνώ. Λέμε για την ανάγκη να δράσουν τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν. Μα η Λευκή Βίβλος υπορίθεται, αν σε όλα αυτά, στην γεωγραφική συνοχή, και καλή θεωρία, αλλά στην πράξη φοβούμαι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ θα ήθελα να φτιάξουμε ένα κείμενο με το οποίο να μην εκφράζουμε μόνο τη λύπη μας για αυτά τα οποία δεν έγιναν. Όταν λέμε για παράδειγμα προσαρμογή, εδώ πρέπει να εμπλέξουμε τις πόλεις, τις περιφέρειες. Γιατί επαναλαμβάνω ωραία θεωρία η εδαφική γεωγραφική συνοχή, αλλά Εδώ έχουμε τις αποδείξεις μπροστά μας για τις επιπτώσεις των επερχομένων αλλαγών. Θα κάνουμε κάτι ή όχι. Φυσικά το κείμενο βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά. Δεν λέμε αρκετά για την εφαρμογή όλων αυτών σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι. Και κλείνουμε λέγοντα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, αλλά είναι, όπως λέμε, ο σαν να περιμένουν οι Γαλοπούλε να έρχονται να έρθουν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τι περιμένετε, τι περιμένουμε. Από πού θα βρούμε τα χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία, από άλλα ταμεία. Δεν μπορούμε εμεί ω Επιτροπή να δίνουμε επιταγή εν λευκό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πιο συγκεκριμένο εξειδικευμένο κείμενο. Κάτι άλλο τώρα. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται αλλαγέ. Γιατί γνωρίζουμε για την αλλαγή του κλίματος, γνωρίζουμε για τις φυσικές καταστροφές που επέρχονται. Έχουμε και το Ταμείο λοιπόν Αλληλεγγύης, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Όμως, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε με τρόπο αρκετά ευέλικτο. Το λέω για να υπενθυμίσω δηλαδή ότι εν μέρη έχουμε επαρκή εργαλεία, μηχανισμούς και κονδύλια για τις δασικέ πυρκαγιέ και το καθεξής. Πληρώνουμε ένα σωρό πόσα για ανατεσώσεις, αλλά συνεχίζουμε να μην είμαστε αρκετά ευέλικτοι. πρέπει στο σημείο αυτό να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις με βάση αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνει το θέμα στη δημοσιότητα, όσο πιο να γίνεται. Πρέπει το κείμενο αυτό να που στη φωνή μας πιο έντονα από οποιοδήποτε άλλο. Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου πιστεύω ότι η συμβολή της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να είναι η εξής. Να πούμε ότι ο αγώνας κατά τη αλλαγή του κλίματο πρέπει να είναι ο κατά προτεραιότητα στόχος μας. Και με βάση αυτό, εν συνεχεία, να δούμε ποια είναι τα εργαλεία. Η μάχη, ο αγώνα δεν γίνεται κατά τομέα, θεματικά αν θέλετε, τομέακα. Χρειαζόμαστε αντιθέτω μια ενιαία πολιτική, συνεπή και συνεκτική, για να αναδιατάξουμε τις εθνικές και τις περιφερειακές μας οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ένα εργαλείο το οποίο όμως απουσιάζει από τις προτάσεις που έχω εδώ μπροστά μου και μιλώ συγκεκριμένα για τα περιφερειακά προγράμματα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Στη Γαλλία συγκεκριμένα έχουμε λάβει μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία την αποκατάσταση δηλαδή, της πολιτικής συνοχής μεταξύ όλων των προσπαθειών περιφερικής ανάπτυξης. Θέλουμε δηλαδή μια περιφερική ανάπτυξη η οποία να μην αντιβαίνει βεβαίως στις ανάγκες που προστάζει η αλλαγή του κλίματος και χρειαζόμαστε φυσικά ε, κάτι για τον τομέα των μεταφορών, της γεωργίας, της πολεοδομίας, της χωροταξίας και του Θα ήθελα λοιπόν τονίσω την ανάγκη τέτοιων αριστείων προγραμμάτων για το κλίμα, ειδικά, τα οποία είναι συμβατά με τα συμπεράσματα της Κοπενχάγης. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στη Λευκή Βίβλο και να αποτελέσει την σπονδυλική στήλη των προσπαθειών μας σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής και τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια κυρίω, όλοι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα τη αλλαγή του κλίματο. Στην χώρα μου, μάλιστα, θα έλεγα ότι το κοινό άρχισε να προσέχει το θέμα λόγω και των τελευταίων πλημμυρών. περιοχέ που δεν είχαν πλημμυρίσει ποτέ πλημμύρισαν τον τελευταίο καιρό και το οποίο κινητοποίησε την κοινή γνώμη. συνειδητοποιούν ότι δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια, είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν και θα ξαναγίνουν. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Η υπερθέρμανση λοιπόν του πλανήτη είναι πλανητικό παγκόσμιο πρόβλημα. Εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι, με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Μερικά από αυτά που ακούστηκαν θέλω να τα σχολιάσω. Το θέμα των ανανεώσιμων πηγών είναι κάτι το οποίο γίνεται όλο και πιο δημοφιλέ, Πολλοί όμω προσπαθούν να μπουν στην αγορά ανανεωσίμων μορφών ενέργεια. παρά το ότι η αγορά δεν είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν εργαλεία και τεχνολογίε που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, μια τεράστια τεχνολογική καθυστέρηση. Και εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Στο τομέα των μεταφορών τώρα. Άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε ένα σωρό εμπόδια. Στους δρόμους και στους σιδηροδρόμους, εμπόδια τα οποία θα συνεχίσουν να προεπλασιάζονται στον εγγύς μέλλον. Βεβαίως, η απόδοση των οχημάτων, των κινητήρων και των οχημάτων βελτιώνεται, αλλά απαιτήθηκαν τεράστιες επενδύσεις και δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν αντίστοιχο των προσδοκιών. Το τι πρέπει να κάνουμε και για τα κτίρια. Τα κτίρια, όπω γνωρίζουμε, είναι υπεύθυνα για το 50% των εκπομπών. Άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα γρήγορα, εάν υπάρχει βεβαίω η πολιτική βουλήση. Και τώρα για τη Γεωργία. Αναφέρθηκε και αυτή. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Η τάση είναι να επιθέμεθα στην Γεωργία, λε και φταίει αυτή από μόνη τη για τι εκπομπέ. Φυσικά έχει μερίδιο ευθύνη όμω. Δεν μπορούμε να τρώσουμε την αξιοπιστία αυτών που δουλεύουν τη γη. Ξεχνώντας για παράδειγμα την βιομηχανία. Κάπου είδα μια αφίσα τις τελευταίες μέρες εδώ στο κοινοβούλιο που λέει ε, λιγότερο κρέα σημαίνει λιγότερη θερμότητα. Δηλαδή να μειώσουμε την παραγωγή κρέατος για να βοηθήσουμε. Ταυτόχρονα όμως ένα δισεκατομμύριο κατοίκων της γης πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε μια μέση οδό, μια λογική μέση οδό. Και τέλος το θέμα τη πυρηνική ενέργεια. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα στην οποία αν αναφέρετε και μόνο την πυρηνική ενέργεια θα σα του βικήσουν ψυχρό στον δρόμο. Λοιπόν, αν περάσουμε το αυλάκι και δούμε την Αγγλία, την Γαλλία, θα δούμε δεκάδες πυρηνικών σταθμών. Η Ευρώπη πρέπει να ιδρύσει μια νέα πολιτική. Να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν μπορούμε να παίρνουμε συναισθηματικές αποφάσεις. Υπάρχει ένα κίνημα και μια τάση στην πυρηνική βιομηχανία υπέρ της ανακύκλωσης των πυρηνικών υποβλήτων. Να δούμε πώς λειτουργεί και να πούμε ένα ναι ή ένα όχι, να ταχθούμε υπέρ ή κατά, μακριά από συναισθηματισμούς. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε μια πολιτική και στον τομέα τη ενέργεια αλλά και στον τομέα τη γεωργία και των μεταφορών. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου ε, ομιλητέ στον κατάλογο. Προθεσμία για κατάθεση των υπολογιών 10 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ συνάδελφοι, σημειώστε αυτή την προθεσμία. Έχουμε μπροστά μα ένα πολύ ενδιαφέροντα στόχο. Πρέπει να αποδείξουμε εδώ τον ρόλο τη περιφερειακή πολιτική στην προσπάθεια αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μας είναι συμβατή με την εν γέννη προσπάθεια και μπορεί να είναι συμβατή και με τις άλλες μελλοντικέ πολιτικές. 10 Δεκεμβρίου λοιπόν, 12 το μεσημέρι. Θα έλεγα να αφήσουμε το σημείο 7 για αύριο, γιατί πρέπει να επιταχύνουμε. Τώρα ξεκινά οι συνεδρία των συντονιστών. Παρακαλώ, όσοι δεν είναι συντονιστές, να αποχωρήσουν. Και θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο στις 9. Παρακαλώ να είστε εδώ στην ώρα σας ακριβής. So, uh, no, uh, um, what I wanted to tell you about the coordinators, yeah, well, studies. Uh, well, you know, the members already read, so you don't have to go for the